<clears throat> Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ε, για την ημερήσια διάταξη, μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη σημερινή μας συνεδρίαση. Έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη και θα καλύψουμε και κάποια γεγονότα της πρόσφατης επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που δεν το συνηθίζουμε ιδιαίτερα. Θα ήθελα γι' αυτό να ευχαριστήσω τους τέσσερις πρεσβευτές της ε, Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας που είναι σήμερα μαζί μας. Ο πρέσβης της Ιταλίας ε, είναι αδιάθετος, δεν θα μπορέσει να έρθει σήμερα εδώ. Έχουμε όμως ε, τον πρεσβευτή της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας και της Ισπανίας. Πρεσβευτές στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας και θα μιλήσουμε μαζί τους για την πρωτοβουλία τη λεγόμενη της Βαϊμάρης. Ξέρετε ότι εδώ και ένα χρόνο περίπου οι υπουργοί του τριγώνου της Βαϊμάρης, δηλαδή από την Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία, απίφθηναν στην ύπατη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μία επιστολή, η οποία επίσης πήγε και στους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ζητούσαν να ξεκινήσει εκ νέου, να δοθεί νέο πνεύμα στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Επικαιροποιήθηκε η πρωτοβουλία αυτή πέρυσι την Άνοιξη και επίσης καλύπτεται και στην έκθεση της κυρίας Άστον, η οποία δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο και η Ισπανία και η Ιταλία στη συνέχεια συντάχθησαν με την πρωτοβουλία αυτή τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να σημειωθεί μια κάποια πρόοδος στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας όσον αφορά το pooling and sharing, και όσον αφορά και την εξέλιξη των θεσμικών αυτών οργάνων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια μιας μόνιμης συνεργασίας σε αμυντικά θέματα. Υπήρξε μια έντονη ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Άστον και την προηγούμενη εβδομάδα οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Υπουργοί Άμυνα συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες και κατέληξαν σε κάποια συμπεράσματα για τα οποία ενδεχομένω να έχετε ενημερωθεί και τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο προφανώς στους τέσσερις ε, πρεσβευτές που είναι μαζί μας. Η εκπρόσωπος της Πολωνίας, η πρέσβης ε, της Πολωνίας θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα του τελευταίου συμβουλίου και ο Γάλλος και ο Γερμανός οι ε, πρεσβευτής θα μπορούσαν να μας μιλήσουν περισσότερο για την πρωτοβουλία της Βαϊμάρης του τριγών της Βαϊμάρης και ο Ισπανός εκπρόσωπος θα μπορούσε να μας εξηγήσει πώς και γιατί οι υπόλοιπες χώρες, συμπεριλαμβανομένης Ιταλίας και της Ισπανίας, έχουν συμπεριληφθεί στην πρωτοβουλία αυτή. Θα εξετάσουμε κατά αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε στο μέλλον από την πρωτοβουλία αυτή. 7-8 λεπτά περίπου ο καθένας, λίγο λιγότερο από 10 λεπτά σας παρακαλώ, προκειμένου να μείνει χρόνος και για τη συζήτηση. Κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο. Euh, Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινησω Έξι 6-8 λεπτά είναι ακόμη περισσότερο από ό,τι αναμέναμε. Μα είχαν πει πέντε αλλά να ξεκινήσω με την εισαγωγή. Να σας πω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας προσκαλέσατε εδώ σε αυτή την Επιτροπή και να σας πω ότι σας είμαστε ευγνώμονες και για την υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια όλου αυτού του έτους και για την υποστήριξή σας σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της ΕΠΑ και την ανάπτυξη και την εφαρμογή της, της πρωτοβουλίας της Βαϊμάρης. Φυσικό δεν μιλάμε μόνο για την ε, ψυχική υποστήριξη αλλά και την υποστήριξη σε είδος ε, γιατί φέτος λάβαμε πολύ σημαντικές εκθέσεις ε, και μια πρόσφατη έκθεση και υπήρχαν και πάρα πολλές συζητήσεις και σεμινάρια και διασκέψεις σε αυτό το βήμα και νομίζω ότι Μας βοηθήσατε με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολύ. Μας δώσατε μεγάλη ορμή. Και μας βοηθήσατε να βελτιώσουμε τις εργασίες μας. Θα μιλήσω και στη μητρική μου γλώσσα. Βλέπω ότι έχω εδώ διερμηνία, αλλά καταρχήν Θέλω να υπογραμμίσω ότι η πρωτοβουλία της Βαϊμάρης όταν ε, αρχίσαμε να τη συζητούμε είχαμε στο παρελθόν ήταν η πρωτοβουλία Χομπίρ το καλοκαίρι του 2009. Ε, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά διέφερε ως οργανισμός ε, και το περιβάλλον εργασίας διέφερε τότε. Δεν είχαμε ακόμα την χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση των θεσμών που ακολούθησε και ακόμη ε, δεν είχαμε τόσες πολλές εξωτερικές προκλήσεις που εμφανίστηκαν ε, φέτος το χειμώνα και την Άνοιξη, με την Αραβική Άνοιξη και τόσες πολλές ε, αλλαγές. Με τις αλλαγές που επισέρχονται στην νότια γειτονιά μας. Όμως ε, ιδέες που παρουσιάζονται από Πολωνία, Γαλλία, Γερμανία ε, ουσιαστικά δημιουργήθηκαν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον ε, και είχαν να κάνουν με διαφορετικές προκλήσεις. Αλλά όπως μας έδειξε η ιστορία, οι ιδέες ε, που συμπεριλάβαμε στην επιστολή ε, της Βαϊμάρης που στην οποία ουσιαστικά αποκρίθηκαν η Ιταλία και η Ισπανία και διάφορες χώρες από διάφορες γωνιές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεμονωμένα κράτη-μέλη. Αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτές οι ιδέες μπορώ να πω ότι εξακολουθούν να ισχύουν, να είναι επίκαιρες. Γιατί, τι μπορώ να πω, ότι για να πετύχουμε τους πολιτικούς μας στόχους για να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας, κυρίως την εξωτερική μας πολιτική, πρέπει να έχουμε τις ε, κατάλληλες ικανότητες ή δυνατότητες. Και φυσικά όλοι βλέπουμε τα οικονομικά προβλήματα, έχουμε περιορισμούς ε, και πρέπει φυσικά να συνενώσουμε τους πόρους μας και να δημιουργήσουμε τους κατάλληλους ε, θεσμικούς μηχανισμούς για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις ιδέες μας και υπάρχει πολιτική βούληση να βρούμε συγκεκριμένους μηχανισμούς και συγκεκριμένες ικανότητες. Αυτό που αναμένουμε στο τέλος ε, του έτους δεν ε, υλοποιήθηκε ε, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ό,τι είχαμε προβλέψει. Ορισμένες ε, ιδέες και πρωτοβουλίες θα, θα τεθούν σε εφαρμογή αργότερα. Όμως ε, η προσοχή μας στράφηκε και σε άλλα προβλήματα. Δεν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε όλα όσα θέλαμε. Αλλά αν δείτε τι συμφωνήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων την 1η Δεκεμβρίου αν δείτε τα σχετικά συμπεράσματα, θα δείτε ότι έχει ξεκινήσει η δουλειά και θα διαρκέσει τουλάχιστον για 6 μήνες. Ε, τουλάχιστον 10 σημεία θα αναφερθούν εδώ, κύρια σημεία των εργασιών μας. Να τεθεί σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα ε, της ανάπτυξης ε, των ε, μη στρατιωτικών ικανοτήτων, έτσι λοιπόν να μπορούμε να ε, αναπτύσσουμε νέες μη στρατιωτικές αποστολές. Έχουμε την ιδέα να ξεκινήσουμε εργασίες για ε, να αναπτύξουμε νέες αποστολές στη Λιβύη, στο κέρας της Αφρικής ε, και στο Σαχέλ. Και επίσης θα αναπτύξουμε στρατιωτικές δυνατότητες και θα θέσουμε σε εφαρμογή πρωτοβουλίες στο ευρύ πεδίο του pooling and sharing σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση πόρων για τις μη στρατιωτικές αποστολές μέχρι τα μέσα του 2012 θα πρέπει να προβούμε σε νέους σχεδιασμούς, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επί νέων διαδικασιών για τη διαχείριση των κρίσεων και κυρίως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την, τον τρόπο επέμβασης ε, σε περίοδους κρίσης ε, και επίσης θα πρέπει να θεωρήσουμε τα έγγραφα που υιοθετήθηκαν κυρίως το 2003 έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα θέσουμε αυτά σε εναρμόνιση με τις σημερινές μας πολιτικές. Και επίσης θα πρέπει να διασύρουμε και τους τρόπους ε, λειτουργίας, σύστασης και λειτουργίας ε, των αποστολών μας επίσης. Ε, αρχίσαμε και εργασίες στο εσωτερικό του επιχειρησιακού κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι το πιο καινούριο καθήκον και θα πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου του 2012, έτσι ώστε να μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή νέε αποστολέ ε, και στα πλαίσια αυτού του επιχειρησιακού κέντρου. Και επίση αποφασίσαμε να συνεργαστούμε πιο στενά με του συνεργάτε μα ε, και να εξεταστούν ε, νέες προτάσεις στις αρχές του 2012. Ίσως να σταματήσω εδώ γιατί ξέρω ότι και οι συνάδελφοι θα σας ε, αναφέρουν πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τις προτάσεις μας, καθώς και θα αναφερθούν και στο ιστορικό της πρωτοβουλίας της Βαϊμάρης, αλλά ήθελα να υπογραμμίσω το εξής. Στην της Πολωνικής Προεδρίας ε, βρισκόμαστε τώρα και τα συμπεράσματα του 2012 δεν ε, ερχόμαστε τώρα στο τέλος της ε, πρωτοβουλίας αυτή. Έχουμε μια ευρεία συνεργασία με πέντε χώρες ε, και έχουμε λάβει κάποιες αποφάσεις, οι οποίες όμως θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή στο μέλλον. Και έχουμε και κάποιες ιδέες που εκκρεμούν. Και φυσικά έχουμε και την ε, αναθεώρηση της ε, στρατηγικής της πολιτικής ασφάλειας και της στρατηγικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πιθανότητα αυτή η αναθεώρηση θα ξεκινήσει του χρόνου. Έτσι λοιπόν έχουμε πολύ μεγάλη πρόκληση ενωπιών μας και είμαι σίγουρη ότι και με τη δική σας υποστήριξη θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή, η συνάδελφος Μπεάτε εξήγησε ποια ήταν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε βρίσκεται στην πολιτική πλευρά των θεμάτων και στα θέματα της άμυνας, όπου τα κράτη-μέλη παραδοσιακά υπενθυμίζουν ότι τα μέσα της πολιτικής αυτής παραμένουν εθνικά μέσα, Νομίζω ότι αν θέλουμε να προχωρήσει το ευρωπαϊκό πολιτικό οικοδόμημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε είναι παρόν στις σχετικές συζητήσεις ε, και πάντοτε θαυμάζω ε, τις θέσεις τις οποίες καταλήγετε στις εκθέσεις σας. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς στο Συμβούλιο να κάνουμε το ίδιο. Εδώ είμαστε μια ομάδα από τέσσερις πρέσβεις και ε, καταρχήν να σας πω ότι για τα αποτελέσματα όλων αυτών εκφράζομαι εξ ονόματος του Συμβουλίου και μάλιστα εδώ ενώπιον του Κοινοβουλίου. Γνωρίζετε ότι σε θέματα ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας η πρωτοβουλία είναι πρωτοβουλία των κρατών μελών και, των υψηλών, και της ΥΠΑ ε, εκπροσώπου. Τα κράτη-μέλη μπορεί να είναι ένα κράτος μέλος, θα μπορούσε να είναι η προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου στη συγκεκριμένη περίπτωση η Πολωνία ή θα μπορούσε να είναι μια ομάδα κρατών μελών. Αυτό είναι το νόημα της πρωτοβουλίας της Βαϊμάρης. Δηλαδή, κατά βάση βρίσκονται τρία κράτη-μέλη, δηλαδή μια ομάδα κρατών μελών, που αποφάσισαν από κοινού να υποβάλουν προτάσεις για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, όπως επιτρέπει η συνθήκη. Υποβάλουν, δηλαδή προτάσεις στο Συμβούλιο και αποφασίζει στη συνέχεια το Συμβούλιο τα χαρακτηριστικά αυτή της ομάδα της Βαϊμάρη ποια είναι. Και να ξεκινήσω από τη Γαλλία, γιατί εγώ από γαλλική σκοπιά τα βλέπω τα πράγματα. Πάντοτε η Γαλλία ενδιαφερόταν για την ευρωπαϊκή άμυνα μέσω της ε, ε, διμερούς διάσκεψης ε, κορυφής το 1998 μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας το 1998 τέθηκαν οι βάσεις. Μετά προχωρήσαμε στη διάσκεψη της Κολονίας αργότερα. Το 2008 φτάσαμε το Δεκέμβριο σε συμπεράσματα ε, τα οποία καθόρισαν σε πολύ ψηλό επίπεδο τις φιλοδοξίες για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας όσον αφορά τις δυνατότητες, ε, τους τρόπους λειτουργίας και επομένως η Γαλλία μέσα σε αυτήν την ομάδα της Βαϊμάρης υπό το ίδιο πνεύμα έχει ενταχθεί. Έτσι βλέπουμε την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. Αυτό είναι το πρίσμα υπό το οποίο βλέπουμε την πρωτοβουλία της Βαϊμάρης και η συνάδελφος Μπεάτε ακριβώς αυτό είπε προηγουμένως. Τον Ιούλιο του 2009 υπήρχε μια πρωτοβουλία μεταξύ του κυρίου Σικόρσκι και του Μπερνάχ Κουσνέ, που ήταν Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας εκείνη την περίοδο, και η Γαλλία σε εκείνη την συνάντηση είπε ότι θέλουμε ένα ισχυρό εταίρο στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και αυτό βλέπουμε στο πρόσωπο της Πολωνίας, μια χώρα που θέλει να προωθήσει το θέμα της άμυνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εμείς θέλουμε να συνοδεύσουμε την Πολωνία σε αυτή την προσπάθειά της και στην καθημερινή μας δουλειά με τη Γερμανία και θα αφήσω το Ιωάννη να μιλήσει για αυτά τα θέματα Θεωρήσαμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της Βαϊμάρης ήταν το κατάλληλο σχήμα για να πάρουν μορφή όλα αυτά, ούτως ώστε να αποτελέσουμε μία ομάδα πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Αυτό που θα ήθελα να πω ε, είναι ότι όσον αφορά τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας, ε, ε, στο Συμβούλιο όλο και περισσότερα κράτη-μέλη από το 2003 και ύστερα Συμμετέχουν σε αποστολές, ευρωπαϊκές αποστολές άμυνας και γνωρίζετε παραδείγματα. Είχαμε 25 τέτοιες αποστολές. Δεν βρισκόμαστε πλέον δηλαδή σε ένα ιδεολογικό ή πολιτικό επίπεδο μόνο, υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα και στην πράξη υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που έχουν πλέον καταλάβει πώς λειτουργούν αυτές οι αποστολές. Όλο και περισσότερα κράτη-μέλη θέλουν να συμμετέχουν και όλο και περισσότερα κράτη-μέλη αντιλαμβάνονται τις ατέλειες του συστήματος και τις δυσκολίες τις οποίες πρέπει να κάνουμε πρόοδο. Και βέβαια η Βαϊμάρη δεν καλύπτει τα πάντα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην πρωτοβουλία της Βαϊμάρης υπάρχουν ε, τρεις πτυχές. Υπάρχει μια πτυχή επιχειρησιακή, όπου θέλουμε να παγιωθούν οι υπάρχουσες επιχειρησιακές δυνατότητες. Υπάρχει μια πτυχή που αφορά τι ικανότητε και άλλη μια πτυχή του πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις ικανότητές μας για την ανάπτυξη μέσων. Για την πτυχή των ικανοτήτων θέλω να πω με σεμνότητα ότι η πρωτοβουλία τη Βαϊμάρη είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε νωρίτερα μέσω του pooling και sharing της συνένωσης και κοινή χρήση που είχε γίνει το Σεπτέμβριο του 2010 στη Γάνδη στην τύπη συνάντηση Υπουργών Άμυνα, όπου και ε, οι Υπουργοί Άμυνα και των 27 κρατών μελών είπαν ότι θέλουν να, αναπτύξουν την ανάπτυξη, να, βοηθήσουν, να προωθήσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων δηλαδή η Βαϊμάρη ξεκίνησε πριν από την σύσταση του τριγώνου της Βαϊμάρης. Τα λέω όλα αυτά για να τονίσω ότι αυτή, αυτό είναι το νόημα της Βαϊμάρης. Είναι ένα σχήμα στο οποίο δεν είναι κατά κανένα τρόπο μόνα τους τα τρία κράτη-μέλη. Και η δουλειά στο τρίγωνο της Βαϊμάρης γίνεται μαζί με την ε, υπηρεσία της ΥΠΑ της εκπροσώπου και μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όλα τα κράτη και τα 27 κράτη υποστηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών την 1η Δεκεμβρίου θέλω να πω ότι η συζήτηση ήταν πολύ δύσκολη ε, γιατί μόλις και ξεφύγαμε από το να μην έχουμε καμία συμφωνία, παρότι πολλά ήταν τα ζητήματα στα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία και τελικά ε, είχαμε, καταλήξαμε στη συμφωνία και χαίρομαι γι' αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο να παρουσιάσουμε τη θέση του Συμβουλίου σήμερα αν δεν είχαμε καταλήξει αυτή τη συμφωνία στη συνάντηση της 1ης Δεκεμβρίου. Χαίρομαι λοιπόν που εμφανίζουμε σήμερα ενώπιόν σα με αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Και υπάρχει τώρα η προοπτική για νέε επιχειρησιακέ δράσει στο κέρα τη Αφρική, στη Λιβύη, στο Σαχέλ Υπάρχει προοπτική της ανάπτυξης δυνατοτήτων ε, μέσω εμβληματικών πρωτοβουλειών, στις οποίες ορισμένα κράτη-μέλη ε, παίζουν τον ηγετικό ρόλο. Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού επιχειρησιακών δράσεων μέσω ε, του κέντρου επιχειρησιακής δράσης και αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν στα τέλη Ιανουαρίου στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και παράλληλα έχουμε και κάποιες μελλοντικέ πρωτοβουλίες. Τον Ιούνιο του 2012 θέλουμε να δούμε τι πρόοδους έχουμε κάνει. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, να βελτιώσουμε τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη που ξεκίνησαν εθελοντικά ε, μετά από μια πρόταση της ε, Πολωνικής Προεδρίας, συνενώθηκαν πολλά άλλα κράτη-μέλη σε αυτή την πρωτοβουλία και τελικά ε, κατέληξαν με ομοφωνία στο Συμβούλιο και των 27 κρατών μελών, κατέληξαν σε αποτελέσματα που ξεκίνησαν από τη Βαϊμάρη, αλλά ξεκινήσαμε τρει και τώρα έχουμε αποτελέσματα των 27 κρατών μελών, πράγμα που είναι πολύ θετικό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Ράιντερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σα ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να λάβω το λόγο σήμερα. Πολλά από αυτά τα οποία θα ήθελα να αναφέρω σήμερα τα είπαν ήδη οι συνάδελφοι. Επομένως ε, δεν θα χρειαστεί ούτε τα 5-6 λεπτά που μας δίνετε να χρησιμοποιήσω. Και θα σας πω περί τίνος ε, πρόκειται. Μιλάμε για την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας ε, που τα λέει όλα. Υπάρχει λέξη κοινή μέσα και μια κοινή πολιτική απαιτεί περισσότερο, κάτι περισσότερο από την πρόσθεση, από το, το άθροισμα των διαφορετικών μεμονωμένων ενδιαφερόντων. Χρειάζεται και ένας προσδιορισμός αυτής της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Και επειδή υπάρχουν περιορισμένοι πόροι, γιατί υπάρχουν ε, δημοσιονομικές πιέσεις, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα σημεία τα οποία μας ενδιαφέρουν και δεν θα πρέπει ο καθένα να ενδιαφέρεται για τα στενά δικά του συμφέροντα. Αυτή η πρωτοβουλία τη Βαϊμάρη προσπαθεί ε, ακριβώς ε, να ελαχιστοποιήσει αυτό το κίνδυνο και να τονίσει το στοιχείο της κοινή πολιτικής, όταν λέμε κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Υπάρχουν δύο σημεία τα οποία έχουμε στην πείρα μας από τις στρατιωτικές ε, και πολιτικές επιχειρήσεις μέχρι τώρα. Πρώτον, ότι χρειαζόμαστε ικανότητα προγραμματισμού και ηγεσία για να μπορέσουμε ε, να βελτιώσουμε ε, τις δράσεις μας και δεύτερον, χρειάζεται να βελτιώσουμε οπωσδήποτε τις συνέργειες η Ευρωπαϊκή Ένωση μας προσφέρει τη δικτύωση μέσω τη οποία μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε και να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη. Το αποτέλεσμα ε, του Συμβουλίου ε, ε, την Πέμπτη που μας πέρασε αποτελεί ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια διαδικασία στην οποία υπάρχουν πολλά βήματα, αλλά είναι μια διαδικασία που έχει τεθεί σε λειτουργία. Και είμαι αισιόδοξο ότι θα μας οδηγήσει σε αυτό το οποίο είχε ως όραμα η πρωτοβουλία της Βαϊμάρης. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρέσβη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα να περιβρίσκομαι απόψε εδώ για να παρουσιάσω αυτές τις ιδέες. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω την ιστορική αναδρομή του Γάλλου συναδέλφου και να σας εξηγήσω γιατί η Ισπανία αλλά και η Ιταλία, ο Ιταλός συνάδελφος ε, δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ σήμερα, Όπω είπε και ο Πρόεδρος, γιατί λοιπόν η Ιταλία και η Ισπανία αποφάσισαν να συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία του τριγώνου της Βαϊμάρη. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, Ισπανική Προεδρία στι αρχέ του 2010, την πρώτη υπό την ε, νέα συνθήκη τη Λισαβόνα σε ισχύ. Εκεί ουσιαστικά εφαρμόσαμε αυτή τη συνθήκη και θέλαμε να υποστηρίξουμε την, υπατορμοστή, συγγνώμη, την εκπρόσωπο ε, για να εφαρμοστεί ε, το περιεχόμενο της συνθήκης. Ε, όμως περιβαλλάνονταν ήδη κάποιες ξεκάθαρες ιδέες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων αμήνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλούσαμε για μια συνέχεια αυτών που, των ικανοτήτων που είχαν παρουσιαστεί από τη Γαλλική Προεδρία το 2008. τότε ε, όταν ε, ανέλαβε την Προεδρία το Βέλγιο, η Βελγική Προεδρία οργάνωσε ε, μια ιδιαίτερα καρποφόρο άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας ε, στη Γάνδη, όπου ανέκυψαν κάποιες ιδέες και το Δεκέμβριο εκείνου του χρόνου οι τρεις χώρες της Βαϊμάρης παρουσίασαν στην ε, πέντε εκπρόσωπο την επιστολή των τριών ή την επιστολή της Βαϊμάρης όπως αποκαλείται. Στην πραγματικότητα η επιστολή αυτή ζητά καταρχήν ε, την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων που προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας ε, στα πλαίσια της ε, ΚΕΠΑ. Δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, ανάπτυξη των, στρατιωτικών και αμυντικών τη ικανοτήτων, ανάπτυξη των θεσμών που περιλαμβάνονται στη συνθήκη τη Λισαβόνα και ουσιαστικά κάτι περισσότερο από την ε, συνέχιση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας. Επίσης, έδωσε όφηση ε, στο οικοδόμημα, στο να δημιουργηθεί ένα οικοδόμημα στον τομέα αυτό και ε, αυτό για να μπορέσει να δοθεί μεγαλύτερη όθηση στην δράση για την θέση εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας η Ισπανία ε, τότε συμφωνούσε πλήρως με τις αρχές αυτές και το ίδιο ίσχυε και για την Ιταλία και ε, είχαμε μια διμερή συνάντηση με τους Ιταλούς συναδέλφους και αποφασίσαμε να στείλουμε μια επιστολή το Μάιο του επόμενου έτους. Ε, αποφασίσαμε να στείλουμε λοιπόν μια επιστολή στην ε, κυρία Άστον και ε, είπαμε ότι συμφωνούσαμε με τις ιδέες αυτές και στείλαμε και ορισμένα έγγραφα όπου αναφερόμασταν σε συγκεκριμένα στοιχεία της Συνδίκλης αγώνας όπως είναι η μόνιμη συνεργασία και η δημιουργία μιας μόνιμης δομής. αυτό ήταν μια συνεισφορά Δείξαμε δηλαδή στου συναδελφού μα ότι μα ενδιαφέρε να συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία τη Βεϊμάρη και στην επόμενη επιστολή που στείλαμε στην Υπατορμοστή, στην το πρόσωπο, με συγχωρείτε. Νομίζω το Μάιο του 2011, όχι, το Σεπτέμβριο του 2011, ε, έχουμε τις πέντε χώρες που υπογράφουν ε, την επιστολή αυτή ε, και υπεγράφει στο ΣΟΠΟΤ ε, στα πλαίσια της άτυπης συνεδρίασης των Υπουργών υπό την Πολωνική Προεδρία. Το τρίγωνο της Βαϊμάρης ε, συγκεντρώνει πέντε χώρες αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνουν αυτές οι πέντε χώρες, το είπε προηγουμένως κάποιος συνάδελφος. Δεν είναι ότι μιλάμε εδώ για ένα περιορισμένο κλαμπ. Ε, ίσως να υπάρχουν πολύ περισσότερα κράτη-μέλη που προσυπογράφουν τις ιδέες αυτές και που θα υποστήριζαν αυτές τις πρωτοβουλίες. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να τονίσουμε ότι αυτές οι πέντε χώρες είναι πέντε από, τις έξι, από τα έξι μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οικονομία, σε πληθυσμό έτσι λοιπόν μιλάμε για πέντε από τα έξι μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν και μεγαλύτερους ε, στρατιωτικούς πόρους που συνεισφέρουν περισσότερο στην άμυνα και έχουν συνεισφέρει περισσότερο ιστορικά στις 25 ε, αποστολές και ΕΠΑ και στρατιωτικές και μη στρατιωτικές. Εκεί έχουν συνεισφέρει λοιπόν περισσότερο και έχουμε και μεγαλύτερες βιομηχανίες άμυνας. Ε, δηλαδή μιλάμε για τις πέντε από τις κυριότερες έξι χώρες αυτή αυτής της ομάδας. Έτσι λοιπόν, εμείς ε, θεωρούμε ότι πληρούμε τις προϋποθέσεις ε, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις ιδέες αυτές ε, και να βοηθήσουμε την κυρία στο να τις αναπτύξει. Γιατί τώρα αυτή η χρονική στιγμή, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, είναι βέβαιο ότι οι προτεραιότητες ανάπτυξης αυτής στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρώθηκαν σε ένα μέσο που ήταν ουσιαστικό για την εργασία της κυρίας Άστον, όπως η ανάπτυξη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Αυτό ήταν αυτή ήταν η δέσμευσή τη και εμεί ε, την υποστηρίξαμε όλα τα κράτη-μέλη. Χρειάστηκε κάποιο χρόνο. Εσεί ε, ξέρετε στο Κοινοβούλιο ποιε ήταν οι δυσκολίε ε, που αντιμετώπισαν η κυρία Άστον και το Συμβούλιο για την ανάπτυξη αυτή τη υπηρεσία. Σήμερα όμω έχουμε μία λειτουργή, έχουμε μία ικανοποιητική υπηρεσία και ω προ το περιεχόμενο και νομίζουμε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να συμπληρώσουμε αυτά τα μέσα. Και εξού οι πρωτοβουλίε αυτές. Το γιατί τώρα. Ποια είναι η σημασία που δίνουμε σε όλα αυτά αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ότι μαζί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση η ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων της ε, Ευρωπαϊκής ε, Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει όλε τι ικανότητε για να μπορέσει να διαδραματίσει ένα παγκόσμιο ρόλο ε, να είναι παγκόσμιος παίκτη, ε, όχι μόνο όπως θέλει το Συμβούλιο, αλλά όπως θέλουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και με αυτό θέλουμε όχι μόνο να δημιουργήσουμε νέους θεσμού, αλλά να μπορέσουμε να δράσουμε. Και αυτό είναι το σημαντικό, να μπορούμε να κάνουμε πράγματα το σημαντικό. Ε, δεν είναι τα νομικά και τα θεσμικά πλαίσια, δεν είναι τα μεγάλα οικοδομήματα, οι μεγάλε δομέ. αλλά μα ενδιαφέρει να μπορούμε να κάνουμε πράγματα από κοινού. Αυτό αναμένει ο κόσμος από την Ευρώπη, αυτό να μένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και αυτό να μένουν οι κύριοι εταίροι της Ευρώπης όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να αναφέρω ένα εταίρο. Και νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε για να απαντήσω και ερωτήσεις ενδεχομένω αργότερα αν υπάρχουν. Ευχαριστώ. merci beaucoup. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις παρεμβάσεις σας αυτές που πραγματικά θέσανε το όλο πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε η πρωτοβουλία αυτή και στο οποίο καταφέραμε να πετύχουμε και τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάσατε. Πρόκειται για αποτελέσματα στα οποία φτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες και έχουν να κάνουν με τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε ομοφωνία ως προς τα εγκριθέντα αυτά συμπεράσματα, μόνο ότι υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις και ακούστηκαν διαφορετικές απόψει κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Από ό,τι φαίνεται όμως ομόφωνα τα 27 κράτη-μέλη ενέκριναν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Πρέπει επίση να πούμε ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα στα πλαίσια τη υποεπιτροπής μα, όσον αφορά την γενικότερη συζήτηση που κάνουμε για την ασφάλεια και την άμυνα, υπάρχει, όπω το είπατε, μια μεγάλη ομοφωνία, μια σημαντική συνένεση, πολλέ διαφορετικέ ευαισθησίε βέβαια, τι οποίε θα συνειδητοποιήσετε στη συνέχεια με τι παρεμβάσει που θα κάνουν οι συνάδελφοι. Σεβόμενοι όμως τις ευαισθησίες αυτές, πρέπει να πούμε, και αυτό αποδείχτηκε πολλές φορές μέσω των εκθέσεων που επεξεργαστήκαμε και που ψηφίσαμε μεγάλη πλειοψηφία στην ε, Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο, και να αναφέρομαι και στον κύριο Γκουαλτιέρη, ο οποίος δυστυχώς απουσιάζει σήμερα, βρίσκεται στη Ρώμη. Έχουμε την έκθεση Γκουαλτιέρη, την έκθεση Λίζεκ, την οποία την οποία θα ψηφίσουμε στην επόμενη σύνοδο της Ολομέλειας. Μέσω των εκθέσεων αυτών φαίνεται ξεκάθαρα ότι ομόφωνα θέλουμε να υποστηρίξουμε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, όχι τόσο από ιδεολογικής πλευράς θα έλεγα, αλλά όπως είπε και ο Ισπανός πρέσβης πριν από λίγο, σε σχέση κυρίως με τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα, τις αποστολές, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να παρέμβουμε επιτόπου έμπρακτα, είτε πρόκειται μέσω μη στρατιωτικών ή ενίοτε στρατιωτικών αποστολών. Ακριβώς λοιπόν αυτή τη δυναμική υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο δυνατόν πιο δυναμικά μέσω αποστολών αξιολόγησης. Ξέρετε ότι για την αποστολή Αταλάντα ήμασταν παρόντες, το ίδιο και για την UTM φέτος. Πρόκειται για μια αποστολή για την κατάρτιση των Σομαλών στρατιωτών. Κάναμε λοιπόν μια έκθεση ανάλυσης και καταφέραμε μέσω αυτής να καταλήξουμε σε κάποιες συστάσεις όσον αφορά την προσαρμογή των αποστολών αυτών και καταφέραμε επίσης να έχουμε και ένα επικοδομητικό διάλογο ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ένα απλό ερώτημα τώρα θα ήθελα να θέσω. Πολλές φορές στα συμπεράσματά σας, τα οποία εγκρίνατε την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρεστε στο νόρο κέντρο επιχειρήσεων. Θα ήθελα ή δυνατόν να μας πείτε τι εννοείται με τον όρο αυτό γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μία ολόκληρη συζήτηση για το κέντρο σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων, αυτό το οποίο ονομάζουμε γενικότερο επιτελείο εμείς πολλές φορές. Επομένως υπάρχουν κάποιες, μια κάποια σημασιολογική σύγχυση ως προς το κέντρο επιχειρήσεων. Αναφερόμαστε στην έκθεση Λίζεξ ότι όντως υπάρχει μια ανάγκη για ένα ουσιαστικό τέτοιο κέντρο σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων για ένα κεντρικό επιτελείο δεν ξέρω αν αναφέρεστε ακριβώς σε αυτό σε συμπεράσματα του Συμβουλίου. Μάλλον σε κάτι εντελώ διαφορετικό αναφέρεστε. Επομένω, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μα εξηγήσετε σε ποια δομή αναφέρεστε, προκειμένου να μην υπάρχει καμία σύγχυση. Έτσι ώστε να μην νομίζει ο κύριο Βανόρντεν ότι προχωρήσαμε πάρα πολύ μακριά ή ότι το Λονδίνο έκανε πάρα πολλέ παραχωρήσει στην έγκριση των συμπερασμάτων. Αυτό είναι το μόνο ερώτημα το οποίο έχω εγώ να θέσω και δίνω το λόγο στον κύριο Λίζε, αντιπρόεδρο της υποεπιτροπή μας και συντάκτη της έκθεσης που θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τον πρόεδρο. Ακούσαμε τις παρεμβάσεις των πρεσβευτών και με έχει καλύψει βέβαια με την ερώτησή του και ο πρόεδρος. Ε, θα ήθελα να κάνω όμως και με τη σειρά μου κάποια άλλα ερωτήματα. Σίγουρα θα ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον να, είναι πολύ ενδιαφέρον να συνομιλούμε με τέσσερις ε, πρεσβευτές. Θα ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρον να είχαμε εδώ και τον Ιταλό πρεσβευτή. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα πιστεύω ότι θα ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρον να μπορούσαμε να είχαμε μαζί μας την Επιτροπή τον πρεσβευτή ή θα έλεγα ακόμα και τον Υπουργό Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου προκειμένου να καταφέρουμε να αλλάξουμε απόψη σε σχέση με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε συζητήσει στα πλαίσια του Κοινοβουλίου μας μέσω των εκθέσεων Ντανζόν, Γουαλτιέρη, μέσω της έκθεσης της δικής μου και θα μπορούσαμε επίση να δούμε ποιε είναι οι επιπτώσει τη χρηματοπιστωτική κρίση στον αμυντικό τομέα. Θα θέλαμε πολύ να γνωρίζουμε ποια είναι η άποψη του Νομένου Βασιλείου σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μου, της σύνταξης της έκθεσής μου, δεν είχα τη δυνατότητα να διαβάσω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ουσιαστικά μόλις πριν από λίγο κατάφερα να τα έχω στα χέρια μου. Καταλήγουμε πάντως εμείς σε κάποια συμπεράσματα στα πλαίσια της δικής μας εισέκθεσης και συμφωνώ απόλυτα με τον πρόεδρο κύριο Ντανζόν. Το EU Operational Headquarters, το κεντρικό αυτό επιχειρήσεων στο οποίο αναφέρεστε, θα ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς ακριβώς παρουσιάζει το Συμβούλιο την γενική αυτή ιδέα και ποια συζήτηση έγινε σε σχέση με αυτό στο Συμβούλιο. Όσον αφορά το pooling and sharing, ένας όρος που χρησιμοποιείται πολύ τελευταία. Νομίζω ότι όλες οι πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τη συνένωση και την κοινή χρήση, με το pooling and sharing και που παρουσιάζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, καταδεικνύουν τελικά ότι η προσέγγιση ουσιαστικά ομοιάζει με τη δική μας την προσέγγιση, παρόλα αυτά κρεμούν ακόμα κάποια ερωτήματα. Γιατί από την εποχή, από την εποχή της επιστολής της Βαϊμάρης μέχρι σήμερα, ελάχιστα πράγματα τελικά ολοκληρώθηκαν. Ακόμα λοιπόν περιμένουμε να ολοκληρωθούν διάφορες πρωτοβουλίες. Επίσης, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου διαβάζει κανείς ότι αναφέρεστε σε μια συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ στα πλαίσια του pooling and sharing. Πολύ ενδιαφέρουσα και η ιδέα αυτή, αλλά υφίστανται κάποιες εμφιβολίες, για παράδειγμα. Σε μερικούς μήνες, σε μερικούς μόλις μήνες, θα έχουμε την Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε να φανταστούμε μια συνεργασία σε αυτό το πλαίσιο δεδομένης της ε, έντασης που υπάρχει μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας. Παρ' όλα αυτά υφίστανται κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ όσον αφορά το κυπριακό ζήτημα. Υφίστανται λοιπόν κάποια ερωτήματα, κάποιες αμφιβολίες, να αναφερθώ σε κάτι ακόμα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός άμυνας. Περιμένουμε πολλά από τον οργανισμό αυτό και στην έκθεσή μας υπογραμμίζουμε την ε, ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξη των ε, δραστηριοτήτων του οργανισμού αυτού, καθώς επίσης και το ότι ο οργανισμός αυτός θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο προπολογισμό. Αν δεν κάνω λάθος, το Συμβούλιο δεν αναφέρεται καθόλου στην κατάρτιση προπολογισμού για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Φαίνεται λοιπόν ότι το Συμβούλιο επιθυμεί να διατηρήσει το status quo. Ουσιαστικά δεν επιθυμεί περισσότερες επιχειρήσεις από τον οργανισμό αυτό. Ευχαριστούμε ο κύριος Πασκού. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του συναδέλφου Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη που δεν μπόρεσε να είναι παρόν σήμερα γιατί έπρεπε ε, ήταν υποχρεωμένος να απουσιάζει και ζήτησε επισταμένος να σας μεταφέρω την συγγνώμη του. Ε, για τα θέματα που συζητάμε υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα του γενικότερου, της γενικότερης έννοιας. Μπορούμε να χωρίσουμε τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη, σε κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, κράτη-μέλη που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης. Αλλά στα θέματα ασφάλειας είναι διαφορετική η κατάσταση. Υπάρχει ένα αίτημα 127 κρατών μελών να θεωρηθεί η ασφάλεια ε, ως κάτι το οποίο αφορά όλους εξίσου. Πώς μπορείτε ε, να ξεπεράσετε αυτή τη δυνητική ε, διάσπαση μεταξύ των δύο επιπέδων. Δεύτερη ερώτηση. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τη δραστική μείωση του στρατιωτικού προϋπολογισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις και ότι πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, αλλά παράλληλα μειώνουμε δραστικά τους προϋπολογισμούς άμυνας. Μιλάμε για ανάπτυξη ικανοτήτων. Με τι χρήματα θα το κάνουμε αυτό αν δεν υπάρχουν χρήματα στον προϋπολογισμό. Και άλλη μια ερώτηση, πώς υπολογίζετε, πώς εκτιμάτε την επιτυχία του τριγώνου της Βαϊμάρης. Θεωρείτε επιτυχία την μείωση των προϋπολογισμών. Ποιοι είναι οι στόχοι ε, του τριγώνου της Βαϊμάρης ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι είναι επιτυχημένη αυτή η προσπάθεια. Και τέλος, όπως είπε ο κύριος Λίζεκ, τι θα γίνει με τη Βρετανία. Έχει ή ο κύριος Βανόρντεν μπορεί να μας έλεγε κάτι τέτοιο. Έχουν εκφράσει κάποιο ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, κύριος Δεφ. Um, I'd like Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση στο Γερμανό πρεσβευτή κυρίω. Το γεγονός ότι η Γερμανία έχει υπογράψει αυτή την επιστολή. Υπονοεί ότι η Γερμανία εφ' εξής έχει αλλάξει τη στάση της στο θέμα της άμυνας και τώρα είναι έτοιμη να διαδραματίσει έναν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη των επιχειρήσεων άμεσα και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ίσως μια ερώτηση προς όλους σας. Ποια είναι τα διδάγματα που προκύπτουν από την επιχείρηση στη Λιβύη. Ευχαριστώ, κύριε Μπραντνερ. Oui, mais, euh, Ευχαριστώ. Deutsch. Θα σας μιλήσω γερμανικά σήμερα. Εδώ υπάρχει μια κατάσταση όπου υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία που αξίζει να τη χαιρετήσουμε έχει δώσει μια όθηση και τώρα έχουμε μάλιστα για κάποια συμπεράσματα και κάποια αποτελέσματα που εν μέρει είναι απογοητευτικά. Είναι θετικό το ότι ξεκινάμε πράγματα, αλλά πού πηγαίνουμε. Μπορούμε να πούμε εντάξει, μια χώρα δεν θέλει να συμμετέχει, να την αφήσουμε στην άκρη και να συνεχίσουμε. Άλλοι πάλι θα πούν ότι δεν πρέπει να το κάνουμε έτσι, αλλά πρέπει όλοι να κινηθούμε μαζί. Νομίζω ότι είναι σημαντικές οι ερωτήσεις. Γιατί μπορούμε να περιμένουμε και άλλα τρία-τέσσερα χρόνια, να περιμένουμε και κάποιες ε, προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπλέον, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας κατά αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε να έχουμε πολιτικέ, μη στρατιωτικέ αποστολέ, τι οποίε δεν χρειαζόμαστε καμία κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Μπορούμε να τα κάνουμε και χωρί κοινή πολιτική άμυνα. Μπορεί να το κάνει η Επιτροπή. Οπότε τι τη χρειαζόμαστε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Εμένα μου λείπει αυτή η βαθύτερη έννοια. Μου λείπει και για το ευρώ, μου λείπει και για το συγκεκριμένο αυτό ε, χώρο της άμυνας. Έχουμε μια εποχή περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε το θάρρος να μιλήσουμε καθαρά και να πούμε ότι θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι σε αυτό το τομέα και ανέφερε και ο κύριος Νταφ τι έγινε ε, με, τη Λιβύη, τι μαθήματα έχουμε, τι διδάγματα έχουμε πάρει. Ε, ε, τι πρέπει να περιμένουμε για να αποκομίσουμε κάποια διδάγματα. Σίγουρα μπορεί ο καθένας να το βλέπει διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι μας ενδιαφέρει να βρούμε απλά συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα μας εξηγήσουν ποιο είναι το βαθύτερο νόημα. Αύριο με το, έχουμε συζητήσεις με το Ινστιτούτο ε, Επιστήμης και Πολιτικής και με την ε, ε, με το ε, Διεθνέ Ίδρυμα Πολιτικής ε, και αύριο ο κύριος Μπιουτικόφερ θα λάβει το λόγο. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίε για συγκεκριμένα προγράμματα και συγκεκριμένα ε, σχέδια. Από τη μια πλευρά κάνουμε μια έκκληση και από την άλλη πλευρά μια παράκληση για μεγαλύτερη ειλικρίνεια και συγκεκριμένα βήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βανόρντεν ήθελε να λάβει το λόγο τήρησα τη σειρά των πολιτικών ομάδων, την αριθμητική σειρά, αλλά ξέρω ότι ε, η δική σας ομιλία θα είναι πολύ πιο πρωτότυπη από τις προηγούμενες, άρα επικάλυψη των ομιλιών δεν διακινδυνεύουμε με τον κύριο Φανόντεν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν να πω στους κυρίους ε, πρέσβεις ε, που μπορώ να πω ότι ότι ε, ήταν σαν να έκαναν ένα χορευτικό και όπως όλα τα χορευτικά το πιο ενδιαφέρον ε, κομμάτι ήταν στο τέλος. Αυτό που είπε ο Ισπανός Πρέσβης ήταν ότι το σημαντικό για την Βεμέρη είναι ότι θα επιτρέψει στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει παγκόσμιο παίκτη και να θέσει σε εφαρμογή όσο επιθυμούν οι πολίτες. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχουμε τους πόρους για να πράξουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι τα είπατε όλα και έχω κάποιες ερωτήσεις για να στραφώ καταρχήν στο Γάλλο πρέσβη. Είπατε ότι η Γαλλία πάντοτε ήταν στραμμένη προς την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ε, φυσικά αν κάτι τέτοιο δεν λειτουργεί, τότε στρέφεστε στο ΝΑΤΟ, όπως είδαμε στη Βοσνία, παραδείγματος χάρη, ή στη Λιβύη. Και εσείς ε, ουσιαστικά ξαναμπήκατε στην ε, ε, διαθρωμένη στρατιωτική δομή της συμμαχίας. Έτσι λοιπόν, να σας ρωτήσω πώς συμφιλιώνεται αυτόν τον προφανή, την προφανή τάση κυριαρχίας του Γάλλου Προέδρου, εθνικής κυριαρχίας του Γάλλου Προέδρου με την αυτό που φαίνεται να παρουσιάζεται εδώ με την επιθυμία δηλαδή για συμμετοχή στις τέτοιες πρωτοβουλίες ε, τώρα να ρωτήσω τον Πολωνό και τον Γερμανό πρέσβη φέρατε τη Λιβύη γιατί δεν ε, βάζετε, κάνετε περισσότερες προσπάθειες ε, για το το μιλήσατε ε, για ολοκλήρωση, αλλά είχαμε το μεγάλο τεστ ε, που ήταν η επιχείρηση στη Λιβύη και να σας πω ότι η Γερμανία ε, πολιτικά και στρατιωτικά και η Πολωνία στρατιωτικά ε, απέτυχαν κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή είχατε πόρους που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Πώς απαντάτε σε αυτό? Και να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι η σημερινή συζήτηση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ολοκλήρωση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ευκαιρία και για μεγαλύτερη ολοκλήρωση στον τομέα της άμυνας. Το βλέπετε δηλαδή αυτό το τμήμα του άλλου. Και να ρωτιέμαι, ποιος ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει σε αυτές τις αποστολές τις οποίες αναφερθήκατε. Μίλησατε για κάποιες φιλοδοξίες τον Ιανουάριο να ξεκινήσουν κάποιες νέες πρωτοβουλίες. Το ιστορικό των αποστολών της ΕΠΑ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε σε άλλους οργανισμούς και τελικά τους κάλεσε να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι. Δηλαδή, Εσεί ε, καταθέσατε το αίτημα τελικά, ζητώντας ευκαιρίες να βάλετε και μια ετικέτα Ευρωπαϊκής Ένωση σε κάποια συγκεκριμένη επιχείρηση. Δεν νομίζω ότι κανένα τράφηκε και σε εσά, ήρθε σε εσά και είπε «Α, εσεί πρέπει να το κάνετε γιατί κανείς άλλο δεν θα το κάνει διαφορετικά». Και κάτι πολύ ενδιαφέρον που έθεσε ο Πρόεδρος μας. Εμένα πραγματικά με συναρπάζει αυτό. Και είναι ο συγκεκριμένο Ε, ορισμός ε, του, του επιχειρησιακού κέντρου. Μπορείτε να μας πείτε πώς ακριβώς διαρθρώνεται το κέντρο αυτό. Ευχαριστώ κύριε Σαγκουράκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να μου επιτρέψετε να εκφράσω μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το πού μας πάτε. Πού μας πάτε ως Επιτροπή και πού μας πάνε οι αξιότιμοι κύριοι ε, πρεσβευτές ε, οι οποίοι πήραν το λόγο σήμερα. Τι εννοώ κύριε Πρόεδρε. Εννοώ ότι βρισκόμαστε σε μια όξυνση των ανταγωνισμών και της αντιπαράθεσης μεταξύ των μεγάλων και των μικρότερων καπιταλιστικών και εμπεριαλιστικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πολύ καλά βιώνουμε αυτή την εποχή, ακόμα όπως θα δούμε και τις επόμενες λίγες μέρες στη Σύνοδο Κορφής στις 9 του Δεκέμβρη. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο ε, Πρεσβευτή από την Ισπανία, τον κύριο Αρίας, διότι έχω την αίσθηση ότι ήταν ο πιο ειλικρινής και ο πιο ξεκάθαρος για το τι τελικά έγινε. Ο κύριος Σαρίας μας είπε την αλήθεια. Δηλαδή, βρέθηκαν οι πέντε πιο ισχυρές καπιταλιστικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές συμφωνήσανε περισσότερο ή λιγότερο σε ένα πλαίσιο και ήρθανε μετά και το επιβάλλαν στους υπόλοιπους 27. Κλασικά πράγματα. Δεν είναι τίποτα καινούριο, δεν είναι τίποτα καταπληκτικό. Το ζήτημα όμως, το απαράδεκτο, είναι να λέγεται ότι αυτό γίνεται στο όνομα των λαών της Ευρώπης. Γιατί ρώτησε κανένας τους λαούς της Ευρώπης ή των διαφόρων χωρών αν θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια στρατιωτική δύναμη επεμβατική και δολοφονική σαν και αυτή που είχε τα τελευταία χρόνια. Δεν νομίζω ότι ρωτήθηκε κανένας γύρω από το ζήτημα αυτό. Και ω εκ τούτου δεν δικαιούται και κανένα να μιλάει εκ μέρους των λαών της Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ένα ζήτημα που εγώ θέλω πολύ συγκεκριμένα να ρωτήσω είναι το εξή. Ωραία, εσεί λέτε βρεθήκατε τρει χώρε οι οποίε ξεκινήσατε μια πρωτοβουλία τη Βαϊμάρη. Πολύ ωραία. Ε, ο κύριο Πρόεδρο τη Επιτροπή είπε ότι τα συμπεράσματα τη Βαϊμάρη είναι συμπεράσματα των 27. Αν κατάλαβα καλά, στι 1 του Δεκέμβρη. Ο κύριος πρέσβης της Ισπανίας μας είπε ότι ακούστε κάτι, είμαστε οι πέντε οι πιο ισχυροί και οι υπόλοιποι θα δούμε τι θα γίνει. Ρωτάω, θα εξακολουθεί να υπάρχει η πρωτοβουλία της Βαϊμάρης ή όχι, από τη στιγμή που υιοθετήθηκε από τους 27. Δεύτερο ερώτημα. Όταν γίνεται λόγος ότι οι πέντε συνοηθήκανε, συνοηθήκανε για τις αμυντικές βιομηχανίες, άρα οι υπόλοιποι 22 θα τις κλείσουν, τι θα κάνουμε. Τρίτο ερώτημα. Διαβάζω σε μια έκθεση της, του Γραφείου Εξοπλισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτό που φαίνεται να υπάρχει περισσότερη κοινή βάση είναι για μη επανδρομένα αεροπλάνα είναι για ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού και είναι για μη επανδρομένα πλοία και νομίζω και για ένα ε, όχημα μεταφοράς προσωπικού. Είναι και αυτό κομμάτι της συμφωνίας της Βαϊμάρης ή αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που υπάρχει. Και τέλος δεν κατάλαβα ποιος ο λόγος για την επιχείρηση στη Λιβύη κύριε Πρόεδρε. Αν θυμάμαι καλά υπήρχε μια απόφαση για αποστολή στρατιωτικής δύναμης Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη στη διάρκεια του πολέμου. Ο πόλεμος τελείωσε Ποιος ο λόγος να υπάρχει ε, αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια διευκρίνηση, αν μου επιτρέπετε, για να είμαστε όλοι σίγουροι ότι μιλάμε για ξεκάθαρα πράγματα. Ο, ο Ισπανός πρέσβης μίλησε για τις πέντε από τις έξι χώρες οι οποίες έχουν τους ε, μεγαλύτερους προϋπολογισμούς στον τομέα της, της άμυνας. Δεν μίλησε για πέντε χώρες απόλυτα, πέντε χώρες που είναι ισχυρότερες και θα επιβάλλουν τη θέση τους στις άλλες. Η πρωτοβουλία της Βαϊμάρης κατέληξε σε ε, ε, συμπεράσματα που υπεγράφησαν από τις 27 χώρες. Επειδή αναφέρετε τις δηλώσεις, ε, την παρέμβαση του Ισπανού πρέσβη, θέλω να τα επαναλάβω, και για την επιχείρηση στη Λιβύη που αναφέραμε, μιλάμε για επιχειρήσεις της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμεσης που μπορεί να είναι μη στρατιωτικές και δεν ξέρω εγώ να αναφέρθηκε αποστολή ε, στρατιωτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λιβύη, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ο κύριος ε, Γιάννης. Ευχαριστώ. Και εμένα μου φαίνεται πολύ σημαντική η διευκρίνησή σας ε, όταν ε, μίλησε ο προηγούμενος ε, συνάδελφος, ε, έβλεπα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου που λέει η Λιβύη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να βοηθήσει τη Λιβύη σε ένα ευρύ πλαίσιο όπως στον τομέα ελέγχου των συνόρων και ελέγχου της ασφάλειας. Από τις αρχές του 2012 θα εκπονηθεί ένα σχέδιο δράσης σεβόμενη τη Λιβυακή κυριαρχία και σε συνεργασία με τον ΟΗΕ. Νομίζω ότι σε αυτό αναφερθήκαν ήταν ε, οι κύριοι πρέσβεις όταν αναφερθήκαν στη Λιβύη, όχι στην ε, επέμβαση απελευθέρωσης του ΝΑΤΟ. Στη Λιβύη ε, η Λιβύη τώρα φυσικά δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωταγωνίστησαν κάποιοι, όχι όλοι, κάποιες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι και μέλη Λοιπόν, φαίνεται και από τις ε, παρεμβάσεις που ακούστηκαν ότι σε αυτό το θέμα έχουμε πάρα πολλές επαναλήψεις γιατί το θέμα της ασφαλείας και της άμυνας φυσικά είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Πάντοτε ήταν. Όμω, πράγματι πρέπει να υπενθυμίσουμε και γι' αυτό λέω ότι πολλέ φορέ κάνουμε επαναλήψει ότι πριν 15 χρόνια ήταν ένα θέμα ταμπού. Δεν μπορούσαμε να το συζητήσουμε υπήρχαν συγκεκριμένε ε, πολιτικέ ομάδε, συγκεκριμένοι βουλευτέ, συγκεκριμένε ε, χώρε που επί τη ουσία καταστούσαν αδύνατο ε, να σημειωθεί κάποιο πρόοδο σε μια πολιτική συνεργασία για να έχουμε κοινή ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο δηλαδή. Δεύτερη παρατήρηση. Πρωτοβουλία τη Βαϊμάρη. Έχει πολύ πρωτότυπε πτυχέ. Κατά την άποψή μου μεταφράζει το ενδιαφέρον τη Πολωνία να προχωρήσει σε μια κοινή ασφαλεία και αμήνα στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι η πρώτη πρωτοβουλία αυτή εδώ. Αναφέρθηκαν και άλλες πρωτοβουλίες από τους κύριους πρεσβευτές που έλαβαν την τελευταία δεκαετία και επίσης ήταν αξιόλογες οι πρωτοβουλίες αυτές. Τώρα, ε, ποιο είναι το μυστικό αυτή τη πρωτοβουλία κατά την άποψή μου, όχι να βελτιωθούν οι στρατιωτικέ στρατιωτικές ικανότητε και δυνατότητε, ε, η υλικοτεχνική υποδομή, οι νομικέ έννοιε ε, αυτών των αποστολών. Απλώ μιλάμε για απαραίτητη όθηση που δίνεται για κάτι πάρα πολύ λεπτό και πάρα πολύ πολύπλοκο που μετρά πάρα πολύ το θέμα τη εθνική κυριαρχία. Αλλά Ορισμένες ε, χώρες και πολλοί βουλευτές είμαστε υπέρ να σημειώσουμε πρόοδο, να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν ε, είναι θετική η πρωτοβουλία της Βαϊμάρης των τριών και κατόπιν πέντε. Μια άλλη παρατήρηση. Το λέω αυτό επειδή ε, ε, άκουσα κάτι που είπε ο προηγούμενο συνάδελφο. Οι πρέσβει ε, ξεκαθάρισαν ότι η πρωτοβουλία τη Βαϊμάρη προτείνει να, μια συμφωνία των πέντε χωρών ε, που αποτελούν τμήμα αυτή, αλλά θα πρέπει φυσικά αυτή η συμφωνία να κυρωθεί από το Συμβούλιο ή θα μετατραπεί σε ενισχυμένη συνεργασία. Σε στην λεγόμενη μόνιμη διαθρωμένη συνεργασία. Όπω τη λέμε τώρα. Και μπορούμε να έχουμε είτε πέντε ή πέντε ακόμα ή τρει ακόμα ή να μείνουν μόνο αυτοί οι πέντε ή το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από ό,τι φαίνεται δεν ε, είναι απαραίτητο να επαναλάβουμε ότι εδώ μιλάμε για κάτι εθελοντικό και ότι οποιοδήποτε μπορεί να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία αυτή όσο υπάρχει ή όταν καταστεί επιχειρησιακή. Τώρα, επόμενη παρατήρηση. Ο κύριος ε, Πάσκου είπε πώς ε, θα τα κάνουμε όλα αυτά με όλο ένα και περισσότερους σπόρους, όλο ένα και περισσότερα χρήματα πριν ε, από την κρίση θέλαμε μια κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας και ακριβώς αν ήταν κοινή, δηλαδή αν σήμερα ήταν απολύτως ενοποιημένη και κοινή θα ήταν πολύ πιο φτηνή. Γιατί δεν θα έπρεπε ε, να συγκεντρώσουμε 27 προϋπολογισμούς ε, και να έχουμε ξεχωριστές πολιτικές, ε, αλλά η ένωση αυτών των προϋπολογισμών ακόμη και σήμερα θα σήμαινε ότι θα είχαμε ένα προϋπολογισμό κατάλληλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως δεν ενώνονται όλοι αυτοί οι προϋπολογιστοί ακόμα. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχουμε και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, και έχουμε και την ε, πολιτική ε, με τους δορυφόρους, ε, έχουμε και τις 25 αποστολές στον κόσμο. Ε, σημειώθηκε πρόοδος, αλλά δεν έχουμε κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, όπως εμένα θα μου άρεσε. Όμως ε, ξέρουμε ότι ε, οι περισσότεροι θα ήθελαν να έχουν μια τέτοια κοινή πολιτική ασφάλειας. Ε, τώρα, για το Ενωμένο Βασίλειο ξέρουμε ε, συνήθως ότι το Ενωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει, ε, όμως ο Μπλερ συμμετείχε στο Σαν Μαλό. Και ίσως μπορούμε να ελπίσουμε ότι ο κύριος Κάμερον θα συμμετέχει σε αυτή σε άλλη πρωτοβουλία που θα υπάρξει σε το θέμα αυτό, γιατί οι κίνδυνοι και οι απειλές είναι κάτι κοινό και ως προς το αποτέλεσμα, δηλαδή στο να υπάρχει συνέχεια, συνέπεια και προβολή, ε, νομίζω ότι αυτά ε, ήδη είναι αποτέλεσμα αυτό καθευτό. Και δεν θα μπω τώρα σε ιστορικά δεδομένα, Νομίζω ότι τώρα και με την πρωτοβουλία της Βημάρης γίνεται μία απόπειρα να εισακάγουμε ε, ουσιαστικά μια Ευρώπη ουσιαστικα από αυτή που είχε από το 1914 στο 1925. Ο κύριος Κάμπελ Μπάνερμαν είναι ο τελευταίος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε τρία σημεία. Πρώτον, την τελευταία φορά που ε, είχε προωθηθεί μια κοινή πολιτική ε, άμυνας για την ε, Ευρώπη, ο τότε υπουργό Σούμαν της Γαλλίας έπρεπε να χρειάστηκε να παρατηθεί. Εγώ είμαι σαφώς κατά ενός κοινού ευρωπαϊκού στρατού και νομίζω ότι προς αυτό ουσιαστικά κινούμαστε τώρα. Δεύτερη ερώτηση. Όσον αφορά τα στρατικά μέσα που θα δώσετε σε, αυτή την, σε αυτή τη στρατιωτική Ευρώπη, πόσα από τα μέσα αυτά έρχονται από το ΝΑΤΟ. Μήπως χρησιμοποιείτε τελικά κυρίως μέσα του ΝΑΤΟ, μέσα που θα χρησιμοποιούσε καλύτερα το ΝΑΤΟ, που θα χρησιμοποιήσετε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ ή ουσιαστικά θα έχουμε νέες ικανότητες, νέα στρατιωτικά μέσα. Τρίτον, προς την πρεσβευτή της Πολωνίας. Ουσιαστικά το ΝΕΤΟ έφερε τη δική σας την ε, ελευθερία. Την ε, εποχή εκείνη που ε, η ε, άστον ουσιαστικά μάζευε περισσότερα χρήματα για την, ε, να προωθήσει τα δικά της ερωτικά συμφέροντα. Για ποιο λόγο εσείς είστε κατά του ΝΑΤΟ. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε πολλές ε, ερωτήσεις. Τώρα, όσον αφορά τις επιλογές του Γάλλου Προέδρου, μπορώ να μιλήσω περισσότερο με τον κύριο Βαν Όρντεν στο Στρασβούργο. Τζέφρι, σε ένα απευθύνομαι όσον αφορά την ε, συνεκτικότητα της πολιτικής του Γάλλου Προέδρου. Ίσως το καλύτερο θα να μιλήσουμε γύρω από ένα γεύμα μαζί στο Στρασβούργο, αν θέλετε. Όχι όμως με έξοδα της Υποεπιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας. Κυρία Πρέσβη, θέλετε εσείς να μιλήσετε πρώτη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα αναφερθώ καταρχάς στην πρώτη ερώτηση που ετέθη από πολλούς παρεμβαίνοντες πρωτοβουλία της Βαϊμάρης και η επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής. Από πού προέρχεται αυτή η πρωτοβουλία και πρόκειται τελικά να δούμε όλα τα κράτη-μέλη να την υποστηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία θα ξεκινήσω και θα ολοκληρώσω ουσιαστικά την παρέμβασή μου λέγοντας ότι τα τρία αυτά κράτη τα οποία έχουν τόσο διαφορετικά ιστορικά χαρακτηριστικά και που έχουν τόσο διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, ακριβώς επειδή αναπτυχθήκαμε εντελώς διαφορετικά ως προς τη δημοκρατία και την οικονομία, σε εντελώς διαφορετικά χρονικά, χρονικές περιόδους. Προκειμένου να καταφέρουν λοιπόν αυτές οι τρεις τόσο διαφορετικές χώρες να μιλήσουν από κοινού για τη δημιουργία μιας κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που μόνο το αποτελεί είναι επίτευγμα. Δεν υπέγραψαν όμως την επιστολή για αυτό το λόγο οι υπουργοί μας. Και ότι για αυτό το λόγο τελικά προτείναμε αυτή την πρωτοβουλία. Προτείναμε αυτή την πρωτοβουλία ακριβώ επειδή έχει κάποιε πολύ συγκεκριμένε ιδέε που έχουν να κάνουν από τη μια με τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, από την άλλη έχουν να κάνουν με την δημιουργία στρατιωτικών ικανοτήτων για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Πρόκειται για ικανότητες διαφορετικές από αυτές του ΝΑΤΟ και το γεγονός ότι η Πολωνία είναι παρούσα στα πλαίσια αυτής της ομάδας ήταν καθοριστικό χάρη στην παρουσία της, προβουλή, της Πολωνίας τελικά τα κράτη-μέλη, 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να συνυπογράψουν αυτή την πρωτοβουλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της πολιτικής άμυνας, ακριβώς επειδή οι αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εντελώ διαφορετικές από τις στρατιωτικές αποστολές του ΝΑΤΟ. Τα δικά μας τα μέσα, οι δικές μας οι αποστολές δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον τομέα της άμυνας, αλλά και με την ανθρωπιστική υποστήριξη, με την ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς επίσης και με τη συνεργασία ανάμεσα στον στρατιωτικό και μη στρατιωτικό τομέα. Ουσιαστικά, η δική μας διαφορα... Ουσιαστικά υπάρχει μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με τον ΝΑΤΟ. Πρέπει κανείς να κάνει μια σαφή διάκριση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει, προσφέρει μέσα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σε, σε περίπτωση εξωτερικής επίθεσης. Είναι περισσότερο μέσα τα οποία έχουν να κάνουν με την σταθεροποίηση κάποιων εξωτερικών ζωνών σταθερότητος. Τα πέντε λοιπόν κράτη της πρωτοβουλίας της Βαϊμάρης συνεργαστήκανε πολύ στενά με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αποκλείστηκε από τη συζήτηση αυτή, από τη διαβούλευση αυτή, κανένα κράτος μέλος. Όλοι συνομίλησαν με όλους και οι υπόλοιποι συναδελφοί μου προφανώς συνομίλησαν με όλους τους συναδέλφους τους στα πλαίσια της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας. Επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για ένα στενό τρίγωνο της Βαϊμάρης για μια ιδιωτική δική μας πρωτοβουλία. Και στο παρελθόν, με την ευκαιρία άλλων συζητήσεων και σε διάφορα φόρα, είχαμε συζητήσει για την πρωτοβουλία της Βαϊμάρης με τους α, συναδέλφους μας από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βλέπετε συμπεράσματα του Συμβουλίου τα βασικά στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας. Και είδαμε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού αποφάσισαν να εγκρίνουν τις ιδέες των πέντε κρατών μελών της Βαϊμάρης ως βάση, ως σημείο εκκίνησης για τις μελλοντικέ μας εργασίες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στα πλαίσια μιας επιτροπής 27 κρατών μελών, προκειμένου από κοινού να εγκρίνουμε περαιτέρω αποφάσεις. Οι προτάσεις της επιστολής της Βαϊμάρης καθώς επίσης και οι πρωτοβουλίες οι οποίες ε, απορρέουν από την επιστολή αυτή ενισχύονται λοιπόν από την υποστήριξη όλων των κρατών μελών γιατί καλούμαστε βέβαια να συνεργαστούμε σε ένα δύσκολο χρηματοοικονομικό πλαίσιο με περιορισμένους προϋπολογισμούς και καλούμαστε να εποφεληθούμε από κοινού από τα περιορισμένα στρατικά μέσα τα οποία διαθέτουμε και να καταφέρουμε από κοινού να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα αυτά για την υπεράσπιση, την άμυνα της Ευρώπης. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποκλείει τη συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ. Το αντίθετο μάλιστα. Όσο περισσότερο είμαστε συντονισμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο περισσότερο θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε και με τον ΝΑΤΟ και θα καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να υποστηρίξουμε καλύτερα και τις αποστολές του ΝΑΤΟ με τα δικά μας τα στρατιωτικά μέσα. Ακούστηκε επίσης ένα ερώτημα το οποίο είχε να κάνει με τη συνεργασία που θα έχουμε με το ΝΑΤΟ στα πλαίσια του pooling and sharing, της συνένωσης και κοινή χρήσης και ποια είναι η τοποθέτηση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε σχέση με αυτό. Κοιτάξτε, επ' αυτού θα συνεργαστούμε με το ΝΑΤΟ προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επικάλυψη και θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε, να αντιγράψουμε τις ε, ιδέες ε, του ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας δεν θα πρέπει να κάνουν τα ίδια πράγματα. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι οι πρωτοβουλίες και οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας θα πρέπει να είναι ευέλικτες, ανοιχτές προς τα έξω να αλληλοσυμπληρώνονται με τις ενέργειες του ΝΑΤΟ και να μην υπάρξει τελικά ένας απόλυτος διαχωρισμός και αποκλεισμός του ΝΑΤΟ από τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολλές οι ερωτήσεις που έχουν γίνει. Ίσως να κάνω μια διάκριση μεταξύ ε, κέντρου επιχειρήσεων ε, και OHQ, γιατί πολλοί από σας κάνατε αυτή την ερώτηση. Υπάρχουν δύο βασικές διαφορές, πιστεύω. Το OHQ δεν υπάρχει. Το κέντρο επιχειρήσεων υπάρχει. Όταν μιλάμε λοιπόν για το κέντρο επιχειρήσεων, δεν μιλάμε για δημιουργία μιας νέας ε, δομής. Μιλάμε για εργασία πάνω στη βάση υφισταμένων δομών. Και αυτό ήταν ε, και αυτό που είπε ο William Hague ε, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών τον Ιούλιο στη μια περίπτωση, σε ορισμένε περιπτώσει, μιλάμε για κάτι το οποίο μπορεί να αποτελεί φιλοδοξία και σε άλλε περιπτώσει μιλάμε για κάτι το οποίο υπάρχει και ομόφωνα το 2004 προσδιορίστηκε από το Συμβούλιο. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο δημιουργεί τη διαφορά είναι ένα επίπεδο φιλοδοξίας και έντασης. Δηλαδή το κέντρο επιχειρήσεων, όπως ορίστηκε το 2004, επιτρέπει να διεξαχθούν κάποιες επιχειρήσεις πολιτικές ή στρατιωτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπει και τη συμμετοχή στον επιχειρησιακό προγραμματισμό αυτών και σχεδιασμό αυτών των αποστολών για τα 27 κράτη-μέλη οι επιχειρήσεις μπορούν να είναι πολιτικές ή στρατιωτικές, αλλά σε επίπεδο έντασης που δεν αντιστοιχεί όμως στο EU Headline Goals, στον στόχο σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης 30.000 στρατιωτών, παραδείγματο χάρη. Υπάρχουν λοιπόν ε, διαφορές και οι συγκεκριμένες ε, ε, περιπτώσεις, οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες θα προσδιοριστούν περισσότερο τον Ιανουάριο ένα άλλο τώρα σημείο που πολλούς ε, σας απογοητεύει, άλλους, ε, δεν για άλλους από εσάς δεν είναι αρκετό. Δεν ξέρω αν το επίπεδο φιλοδοξίας μας είναι υψηλό. Πάντως αυτό το οποίο θέλουμε είναι να συνεχίσουμε ε, τις εργασίες μας και μάλιστα ομόφωνα σε αυτό το θέμα. Και η επιτυχία της διάσκεψης του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου, επιτυχία εντός εισαγωγικών, είναι ότι μέσα σε ένα επίπεδο πολύ σοβαρής οικονομικής κρίσης, βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη διατηρούν ένα επίπεδο φιλοδοξίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που έχουμε ε, πολιτικές κρίσεις στο κέρας της Αφρικής, στο Σαχέλ, στη Λιβύη δυνητικά, και δεύτερον, και εδώ απαντώ και στον κύριο Βαν Όρντεν για το, το ότι δεν υπάρχει κάτι πραγματικά συγκεκριμένο, δηλαδή η ιδέα του ότι χανόμαστε σε θεσμικό επίπεδο και δεν κάνουμε τίποτα συγκεκριμένο. Θα έλεγα διαβάστε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Υπάρχει απόφαση να ξεκινήσουν κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα, ευρωπαϊκά έργα για την ανάπτυξη ικανοτήτων, δηλαδή σε αυτά θα συμμετάσχουν κράτη-μέλη που έχουν δηλώσει τη θέση τους για τη δυνατότητα ε, εκπαίδευσης ε, πιλότων μαχητικών αεροσκαφών, για τη δυνατότητα παροχής βοήθειας ε, και ιατρικής βοήθειας. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες φιλοδοξίες. Όλα αυτά δεν μας εμποδίζουν να βελτιώνουμε την ικανότητά μας για σχεδιασμό χρησιμοποιώντας το εφιστάμενο κέντρο επιχειρήσεων. Για αυτό το οποίο ρώτησε ο κύριος Νταφ ε, για τα διδάγματα από τη Λιβύη, ένα πρώτο δίδαγμα είναι ότι οι Ευρωπαίοι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ δεν είχαν ικανότητες ε, και γι' αυτό έγιναν οι προσπάθειες ε, να παρασχεθεί αυτή η απάντηση, όπως σας είπα. Και δεύτερον, δεν είχαμε δυνατότητα αντίδρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά ε, ε, την απόκριση στρατιωτικών δράσεων και το κέντρο επιχειρήσεων μπορεί να προγραμματίσει κάποιες επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο δίνει μία αρχή ε, απαντήσεων, μια, κάποια πρώτη απάντηση. Δεν συμφωνώ στη συνέχεια απολύτως με αυτά που είπε η κυρία Μπρόντνερ δεν εγκαταλείπουμε την, ευρωπαϊκή, κοινή πολιτική ασφάλειας, την πολιτική και άμυνας. Υπάρχει μια υπεραξία που είναι ίσως περισσότερο πολιτική, περισσότερο στοχευμένη και που εμπλέκει περισσότερο το Συμβούλιο, είναι περισσότερο ορατή και μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον στοιχείο απάντησης στην περίοδο κρίσης. Ο κύριος Βανόρντεν ανέφερε τις στρατηγικές επιλογές της Γαλλίας, σας παραπέμπω στις ομιλίες του Πρόεδρου της Δημοκρασίας. Υπάρχει μια λευκή βίβλος του 2008 που κατευθύνθη κατόπιν αιτήματος του Νικολά Σαρκοζή, όπου αναγράφεται ότι η Γαλλία παραμένει πλήρως δεσμευμένη και υπάρχουν διάφορα στοιχεία που αφορούν τη Γαλλία και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής άμυνας. Η πλήρη συμμετοχή της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ, θέλω να πω ότι ε, πάντοτε τόνιζε η Γαλλία ότι δεν ε, είναι άσχετη από την βούλησή μας να αναπτύξουμε μια ευρωπαϊκή άμυνα και δεν υπάρχει απουσία βούληση συμμετοχής στο ΝΑΤΟ. Θελήσαμε να δείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε παρόντες και στους δύο οργανισμούς. Και σας παραπέμπω και πάλι σε όλες τις ομιλίες του Γάλλου Προέδρου για να σας αποδείξω ότι η Γαλλία δεν εγκατέλειψε αυτή τη φιλοδοξία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αρχίζει επιχειρήσεις ε, κατόπιν ετήματος. Δεν ξεκινάμε εμείς με τις αποστολές. Μας υποβάλλεται κάποια, κάποιο αίτημα και αν ε, βρισκόμαστε στη Λιβύη, βρισκόμαστε σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο κατόπιν ετήματος που μας απευθύνθηκε. Ο κύριος Καμερμπένεμαν μας ρώτησε αν θα λάβουμε πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες δεν ανήκουν ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πρωτοβουλίες ανήκουν στα κράτη-μέλη, στους συμμάχους, στο ΝΑΤΟ. Και στη συνέχεια τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφασίσουν εάν ε, θα συμμετάσχουν σε αποστολές των ε, ένα ή στον άλλο οργανισμό. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι και βέβαια έχει λόγο ύπαρξης η, Ευρωπαϊ... η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και αυτό είναι θέμα και πολιτικών επιλογών και κάθε φορά ποικίλουν οι ετούντες, ποικίλει ο χώρος στο οποίο διεξάγεται μια αποστολή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει η η κοινη πολιτικη Ένωση και αμυνα και αυτο ειναι θεμα και πολιτικων επιλογων και καθε φορα ποικιλουν οι ετουντε ποικιλει ο χωρος στο οποιο διεξαγεται μια αποστολη υπαρχουν πραγματα τα οποια μπορει να κανει η ευρωπαικη ενωση και οχι το ΝΑΤΟ και δεν υπάρχει αντινομία μεταξύ των δύο. Εάν αναπτύσσουμε δυνατότητε στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αφαιρούμε κάτι από το ΝΑΤΟ. Είναι απόφαση των κρατών μελών που θα αποφασίσουν τι θα κάνουν τελικά. Ευχαριστώ. Ο Γερμανό Πρόεδρο έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε εδώ οι πρέσβεις από το τρίγωνο της Βαϊμάρης και ο Ισπανός συνάδελφος, αλλά εδώ μιλάμε για μια κοινή απόφαση που έλαβαν τα 27 κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για μια πρωτοβουλία της Βαϊμάρης, γιατί στο μεταξύ υπάρχει συνένεση. Είναι μια απόφαση του Συμβουλίου που ελήφθη με συνένεση των 27 κρατών μελών. Αυτή η απόφαση του Συμβουλίου δεν αποτελεί επικάλυψη, ούτε ανταγωνίζεται το ΝΑΤΟ προχωρεί προς την κατεύθυνση της ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ε, που ακριβώς ε, αποτελεί μια λύση σε περιπτώσεις μικρότερης έντασης όπου το ΝΑΤΟ είτε δεν ενδιαφέρεται είτε δεν έχει τα κατάλληλα μέσα. Αν παραδείγματο χάρη δούμε την εκπαίδευση της αστυνομία στο Αφγανιστάν ή αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γεωργία. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα καθήκοντα που μπορεί να εκπληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση άριστα. Μέσω της απόφασης του Συμβουλίου δεν μιλάμε για πόρους του ΝΑΤΟ και όπως είπε πολύ σωστά ο, συνάδελφος, ο Γάλλος συνάδελφος, οι πόροι ή τα μέσα είναι μέσα των κρατών μελών και τα κράτη-μέλη αποφασίζουν ανά αποστολή, ανά συγκεκριμένη πρόκληση, ε, ε, τι επιχείρηση πρέπει να αναλυθεί. Και εδώ υπάρχει το pooling and ε, sharing που δεν ε, βρίσκεται σε ανταγωνιστική θέση. Χέρι με χέρι βαδίζουμε με τον ΝΑΤΟ και συνεργαζόμαστε σε αυτά τα θέματα. Όσον αφορά την εμπλοκή της Γερμανίας, ε, για την οποία με, ρωτήσατε κύριε Βουλευτά, η Γερμανία είναι μία από τις πολύ λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, έχει συμμετάσχει σε όλες στις αποστολές της ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και στο Κωσυφοπέδιο και στο Αφγανιστάν στο Αταλάντα και έχουμε και το κέντρο δράσεων εκεί. Επομένως, ε, δεν νομίζω ότι τα σχόλια αυτά είναι απόλυτα εύστοχα. Για την επιχείρηση στη Λιβύη δεν θέλω να επεκταθώ γιατί νομίζω ότι θα μας ε, κάνει να παρεκκλίνουμε από το θέμα μας. Είμαστε όμως έτοιμοι και αν ε, τεθεί το θέμα αποστολής στη Λιβύη θα υπάρξει κατάλληλη απάντηση και δεν νομίζω ότι ε, έχει φτάσει στο τέλος της ε, αποτυχάνει η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε την Πέμπτη με συνεργασία των 27 κρατών μελών θεωρώ ότι είναι πραγματική επιτυχία. Και αυτή η απόφαση του Συμβουλίου θέτει σε λειτουργία ε, μια διαδικασία που στα τέλη Ιανουαρίου θα πρέπει να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα Μπορεί να, είναι να μιλάμε για αποστολή στο κέρα της ε, Αφρικής ή κάτι άλλο. Αλλά αυτό το οποίο θα είναι στο τέλος της διαδικασίας δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να προδικάσουμε από τώρα. Νομίζω ότι θα ήταν σφάλμα το να κλείσουμε τώρα την πόρτα σε αυτή τη συμμετοχή όλων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει κάπως με τον χρόνο, αλλά ήθελα να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις ορισμένοι από εσάς αναφερθήκατε σε αυτές τις εξελίξεις ε, τη στιγμή που υπάρχει μείωση των προπολογισμών για την άμυνα στην Ευρώπη. Ακριβώς για το λόγο αυτό τα σχέδια τα οποία μιλήσαμε και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτή τη στιγμή αυτό το pooling and sharing συνένωση και κοινή χρήση. Δηλαδή δεν μιλάμε για να έχουμε μεγαλύτερο προπολογισμό, αλλά να το χρησιμοποιήσουμε τον προπολογισμό που έχουμε με πιο εξορθολογιστικό τρόπο. Πιο ορθολογιστικό τρόπο. Ε, σύμφωνα με την ε, ε, Επιτροπή, Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φτάνουμε σήμερα στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ε, ως προϋπολογισμό προπολογισμό των 27, δηλαδή μιλάμε τα δύο τρίτα του προπολογισμού των ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα έχουμε παρόμοιο ε, αριθμό με τους προπολογισμούς Κίνας, Ιαπωνίας, ε, ε, Ρωσίας, Κίνας, Σαουδικής Αραβίας από κοινού. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να απτύξουμε αυτή τη συνεργασία για να, για να χρησιμοποιήσουμε ε, καλά αυτό το προπολογισμού. Έχουμε ένα εκατομμύριο, 700.000 στρατιώτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως ένα πολύ μικρό τμήμα αυτών αναπτύσσονται στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αν χρησιμοποιούνται καλά, ε, τα στρατεύματά μας. Ε, και ο κύριος Βανόρντεν ε, αναφερθήκατε, αναφέρθηκε στο αν έχει νόημα μια πολιτική αμυνάς. Ε, φυσικά και έχει νόημα ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να διαδραματίσει παγκόσμιο ρόλο αν δεν έχει μια αξιόπιστη πολιτική στον τομέα της ασφαλείας και της άμυνας. Και, και σε σχέση ε, με τους Ευρωπαίους πολίτες, κοιτάξτε, εγώ είπα ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες στην πλειοψηφία τους θέλουν κάτι τέτοιο και ίσως ε, να απαντήσω. Άκουσα πολύ προσοχή τι είπε ο κύριος Αγκουράκης, ε, ο οποίος ανέφερε ε, αρθήκε σε δύο ρήματα που πραγματικά τραβήξαν την προσοχή μου. Εγώ δυστυχώς ε, θεωρώ ότι πολύ λίγο ακούω τις Βρυξέλλε και πάντα επιβάλλω και σκοτώνω. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ μακριά από τις ε, θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Δεν νομίζω ότι θέλουμε εδώ να επεμβαίνουμε και να σκοτώνουμε. απλώ θέλουμε να σώζουμε ζωές και να προστατεύουμε τη ζωή. Και εγώ νομίζω ότι σε αυτή τη συνένωση, με αυτό το pooling, ε, δεν θέλουμε εδώ τα πλέον εκτήματα των πέντε ε, βιομηχανιών. Θέλουμε όλες οι βιομηχανίες όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, να υποφεληθούν ε, καλύτερα από τις επενδύσεις τους. Έτσι, λοιπόν, το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχο έχουν να προστατεύουν την ειρήνη και να τη διατηρούν. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία λοιπόν κυρίες και κύριοι πρεσβευτές. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Θα έχουμε τη δυνατότητα στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια, την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την κυρία Άστον. Θα επανέλθουμε λοιπόν στα ζητήματα αυτά και στα συμπεράσματα τα οποία συζητήσαμε. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής συνεδρίασης. Θα μιλήσουμε με την κυρία Κλόντ Αγνού και με τον στρατηγό Στεφάν Αμπριάλ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν παρόντες ε, στην υποεπιτροπή μας και είμαστε στην διάθεσή σας προκειμένου να συνεχίσουμε τον ε, μεταξύ διάλογο. Το είπατε και εσείς στα συμπεράσματα της προηγούμενης εβδομάδας. Ήδη προβλέπετε ένα ραντεβού σημαντικό τον Ιανουάριο, προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί το Κέντρο Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι σημαντικό να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πρωτοβουλία αυτή. Μας ενδιαφέρει και εμάς ιδιαίτερα. Είδατε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα ευαισθησιών σε τα πλαίσια αυτής της υποεπιτροπής, σε κάθε πάντως περίπτωση θα πρέπει τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο και όσον αφορά τις στρατιωτικές ικανότητες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις αποφάσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται και από τους 27. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και βέβαια ο Βρετανός σας συνάδελφος μπορεί και αυτός να έρθει όποτε θέλει και να μας μιλήσει για τα ζητήματα αυτά. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Καθίστε παρακαλώ πολύ. Έχω την ευχαρίστηση να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας δύο ανθρώπους που έρχονται συχνά στην υποεπιτροπή μας την Claude France αρνού, εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα και τον στρατηγό Στεφάν Αμπριάλ, ανώτατο συμμαχικό διοικητή μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ στι Ηνωμένε Πολιτείε, ο οποίος μας κάνει ιδιαίτερη, ιδιαίτερη τιμή με την πολύ συχνή παρουσία του εδώ. Κάθε φορά που έρχεται θα έλεγα, αλλά όχι, ξέρω ότι έρχεστε πολύ συχνά στην ε, Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε πολύ που έρχεστε συχνά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιλήσαμε με τους πρεσβευτές του τριγώνου της Βαϊμάρης που συμμετέχουν στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας τις πρωτοβουλίες του όσον αφορά την ε, κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, ιδίως στα πλαίσια της ε, συνένωσης και της κοινή χρήσης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο διαδικασίες αυτή τη στιγμή οι διαδικασίες pooling and sharing, όπως λέμε και στα γαλλικά λέει ο πρόεδρος, και της smart defense, της εφίους άμυνας, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ αυτή τη φορά όμως. Και κάθε φορά προσπαθούμε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή σύγκληση στις ε, πρωτοβουλίες ε, στις οποίες προχωρούν οι δύο αυτοί οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, Σύγκληση που είναι πολύ σημαντική, ιδίω σε μια περίοδο χρηματοπιστωτική κρίση όπου συρρυκνώνονται οι αμυντικοί προπολογισμοί. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να επιμεριστούμε κάποιε στρατιωτικέ μα ικανότητε. Προτού μιλήσουμε για την κοινή αυτή συνεργασία που συναντά κάποια θεσμικά και πολιτικά προβλήματα και τα οποία τα γνωρίζουμε, θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο σας απασχολεί πολύ συχνά και τους δυο σας, το να καταφέρετε δηλαδή να εντοπίσετε τις ε, δυσκολίες αυτές που υπάρχουν στη συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε φορά που καλούνται να επιτελέσουν μια κοινή εργασία. Θα θέλω λοιπόν να γνωρίζουμε και εμείς πώς έχουν τα πράγματα, να μας πείτε ο καθένας στον οργανισμό σας, αλλά και από κοινού, ποια είναι τα σημεία εκείνα τα οποία θεωρείται ότι θα, στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα πλαίσια του κοινού επιμερισμού, ποιε είναι όμως και οι δυσκολίες οι οποίες παραμένουν τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, δυσκολίες που θα πρέπει να ξεπεράσουμε προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια αποτελεσματική κοινή χρήση των δυνατοτήτων μας. Ο κύριος ε, Αμπριάλ θα μπορούσε να μας μιλήσει και για την προετοιμασία της Συνόδου του Σικάγο. Τι μπορούμε να περιμένουμε από τη Σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ την ερχόμενη Άνοιξη. Σας δίνω ευθύ αμέσω το λόγο. Η κυρία Αγνού θα μας μιλήσει ε, προσωπώντας τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πραγματική τιμή μου να παρευρίσκομαι εδώ σήμερα. Για μας ε, ήταν ε, πάρα πολύ σημαντική στιγμή όταν η Επιτροπή σας για την Ασφαλεία και την ε, Άμυνα επισκέφθηκε τον οργανισμό μας. Για μας είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε πόσο ενδιαφέρεστε και συνεχίζει χωρίς μικρόφωνο η μιλήτρια. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε μια συζήτηση για τόσο πράττουμε. Τώρα βρισκόμαστε τρει-τέσσερι ημέρε μετά την ε, Σύνοδο των Υπουργών Άμυνα, 30 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο φυσικά του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά και στο πλαίσιο τη ε, Διεθνήνουσα Επιτροπή ε, του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα. Και θα ξεκινήσω από εκεί, γιατί νομίζω ότι αυτό σημείωσε ένα σημαντικό στάδιο, ένα νέο στάδιο για το pooling and sharing, συνένωση και κοινή χρήση χρήσης. πολύ sharing. Και πραγματικά νομίζω ότι έτσι περνάμε από τη θεωρία στην πράξη και βρισκόμαστε έξι μήνες μετά από την εντολή των Υπουργών Άμυνα που δόθηκε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα τον περασμένο Μάιο και τα αποτελέσματα ήταν υποσχόμενα γιατί είχαμε ε, πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή σημειώνεται ένα πρώτο στάδιο ενώψη μια μιας που θα επιτρέψει να πάμε ε, παραπέρα. 11 σχέδια τέθηκαν, ε, υποφελήθηκαν στα κράτη-μέλη και ε, τοποθετήθηκαν θετικά όλοι οι υπουργοί που πήραν το λόγο και μπορώ να σας πω ότι τελικά καταλήξαμε σε 13 ε, σχέδια γιατί κάποιοι υπουργοί πρόσθεσαν κάποιες προτάσεις και έτσι λοιπόν αυξήθηκε ο κατάλογος των όσων είχαν υποβληθεί βάσει των συγκεκριμένων δεσμεύσεων και ε, για μια ακόμη φορά πρόκειται για συγκεκριμένε δεσμεύσει ε, και ε, αυτό από τα περισσότερα κράτη-μέλη που ουσιαστικά λαμβάνουν έναν ηγετικό ρόλο ε, για τις διάφορες ε, ικανότητες ε, ή ηγετικό ρόλο στη συμμετοχή. Ορισμένα παραδείγματα αυτών συγκεκριμένων δεσμεύσεων σε ό,τι αφορά την κοινή μονάδα επικοινωνιών μέσω δορυφόρων. Έχουμε έξι κρατημέλη που ζήτησαν να συμμετάσχουν πέρα από αυτούς που έχουν ήδη υπογράψει σε ό,τι αφορά τον ιατρικό γεωργικό κλάδο. Εκεί ε, έχουμε έξι κράτη-μέλη που δήλωσαν την υποστήριξή τους ε, και με ένα κράτος Ιταλία που δήλωσε ότι είναι έτοιμο να αναλάβει τη διεύθυνση των εργασιών. Αυτό για να υποστηρίζονται οι στρατιώτες μας ε, στο θέατρο. Ε, των επιχειρήσεων και να σας πω ότι η Ιρλανδία θα αναλάβει τις εργασίες ε, της κατάρτισης ε, στον ναυτικό τομέα, η Ιταλία για τα ιατρικά και για την κατάρτιση των πιλότων και η Γαλλία για την κατάρτιση των πιλότων μεταφοράς. Η Ιταλία δηλαδή επικεντρώνεται περισσότερο στους πιλότους των καταδιοκτικών και η Φιλανδία συνεχίζει ήδη τις πολύ προχωρημένες εργασίες για την εποπτεία στην ε, θάλασσα. Ε, οι ικανότητε ε, αυτές ήταν ουσιαστικές για να ενισχυθεί και η αυτόνομη ικανότητα δράση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτοντας ορισμένα από τα κοινά που είχαν ανακύψει στην επιχείρηση της Λεβής, τον ανεφοδιασμό, παραδείγματο χάρη, τα μέσα αναγνώρισης ε, και εποπτείας και παρακολούθησης και όπως ξέρετε οι Ηνωμένε Πολιτείε είπαν πολύ ξεκάθαρα ε, και σε ένα λόγο τον κύριο Γκέτση και στον κύριο Πανέτα ότι δεν ήταν διατεθειμένες ε, να δρουν στη θέση των Ευρωπαίων και ότι έπρεπε οι Ευρωπαίοι να είναι σε θέση να αναπτύσσουν αυτές τις ικανότητες για τέτοιες επιχειρήσεις. Και επίσης, ε, Τώρα, όπως σας είπα, έχουμε και την ιατρική υποστήριξη, το θέμα των μεταφορών και επίσης να έχουμε ε, και ε, πληρώματα που να μπορούν να αναπτυχθούν και επίση να βελτιώσουμε τη δυνατότητα ανάπτυξης των ευρωπαϊκών ικανοτήτων ή δυνατοτήτων. Την ε, περασμένη εβδομάδα λοιπόν έγινε ένα πρώτο βήμα με αυτό το pooling and sharing που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Θα αναφερθώ στο παράδειγμα ε, των ε, δορυφορικών επικοινωνιών. Η ε, μονάδα εφοδιασμού επικοινωνίας μέσω δορυφόρου είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσω μόλις το χρειάζονται τα κράτη. Από την άλλη εργαζόμαστε σε μια πιο συστηματική προσέγγιση για να προετοιμάσουμε το μέλλον, δηλαδή από τη στιγμή της έγκρισης όσον ε, ε, όσων συζητήθηκαν την ε, περασμένη εβδομάδα και επίση, λαμβάνοντα τη σκητάλη όσων ήδη λειτουργούν στο pooling and sharing και να δούμε υπό ποιες πιο προθέσει. Ο στόχο μα λοιπόν ήταν να δείξουμε πόσο σκόπιμη είναι η έννοια αυτή, να αρχίσουμε να δημιουργούμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, γιατί αυτό αποτελεί στοιχείο κλειδί ε, δεν μπορούμε να συνενώσουμε και να έχουμε κοινή χρέση αν ε, δεν υπάρχει αμοιβή εμπιστοσύνη. Και φυσικά πρέπει να έχουμε και ψυχολογική εμπιστοσύνη, αλλά θα πρέπει να έχουμε και τις κατάλληλες ρήτρε για να μπορέσουμε να προβούμε σε αυτή την συνένωση για να χρησιμοποιήσουμε από κοινού αυτές τις ικανότητες ξέρετε ότι είχαμε και το διαγωνισμό προσωπικού του ψηλοπιπέδου. είχαμε τους ε, ε πρώην ε, του Γενικού Επιτελείου της ε, Ιταλίας, ο κ. Πλωνίου και Σιρό και είχαμε και τον στρατηγό Ματνίτσον από τη Σουηδία και το σημερινό Φιλανδό επικεφαλής εξοπλισμών. Και με τη Σουνσοράμ... Ε, του Φιλμαρινέκα και αυτό μας επέτρεψε να μεταβούμε στις πρωτεύουσες και να επιβεβαιώσουμε ποιες είναι ε, οι προϋποθέσεις ε, για να περάσουμε στο pooling and sharing στην πράξη και να δούμε ε, τι γίνεται με την εθνική κυριαρχία και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητες που έχουμε στη διάθεσή μας, να δούμε και τι ισχύει στη βιομηχανία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υποστηρίξουμε τη συνένωση και την κοινή χρήση κυρίως στο δύσκολο πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε και επίσης να έχουμε και βιομηχανικές και τεχνολογικές αιστείες. Και έχουμε και το χρηματοοικονομικό ζήτημα. Επικεντρωθήκαμε πολύ σε αποστολές υποστήριξης γιατί ε, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα Υπουργεία Αμυνάς μας θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από δράσεις που δεν μας ε, ζητούν πολύ σημαντικές επενδύσεις γιατί θα ήταν κάτι μη ρεαλιστικό. Έτσι λοιπόν ε, επικεντρωθήκαμε σε όσα μπορούν να γίνουν αμέσως με την ελπίδα ότι ε, κάνοντας τέτοιες οικονομίες αυτό θα πέτρεπε στα κράτη-μέλη να επικεντρωθούν σε δεύτερο χρόνο σε πιο μακροπρόθεσμες δράσεις και ε, σε προγράμματα απόκτησης και έρευνας στον τεχνολογικό τομέα. Δεύτερο στοιχείο κλειδί, ότι αφορά τεχνικά, νομικά ε, ζητήματα για να θέσουμε σε εφαρμογή αυτή τη συνεργασία. Είδαμε ότι έχουμε κάποιες συνεργασίες που λειτουργούν πολύ καλά και κυρίως ε, μιλάμε για περιφερειακές συνεργασίες που λειτουργούν ε, πολύ καλά, ότι ο ένας μπορεί να μάθει από τον άλλο και νομίζω αυτό είναι και το ενδιαφέρον αυτού του εγχειρήματο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές και με κανονιστικούς και νομικούς όρους ε, και οικονομικού όρους έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει μια συνεργασία και να πράξουμε έτσι ώστε να έχουμε μια καθολική εικόνα των συνεργασιών αυτών για να μπορούν να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και τα κρατημέλη για όσα θέλουν να κάνουν από κοινά, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια διαφάνεια ε, και να δούμε αν μέσω αυτής της συνεργασίας αν καλύπτουμε κενά ικανοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή αν αντίθετα δημιουργούμε υπερβολικές ικανότητες σε ορισμένο τομέα, σε ορισμένους τομείς αφήνοντας τρύπε κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν ε, και πάλι σεβόμενη την απόλυτη κυριαρχία των αποφάσεων αυτών θα πρέπει ε, να έχουμε μια καθολική εικόνα του εγχειρήματο σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την διαχείριση και την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων. Η πρόθεσή μας μας είναι βάση της στήριξης των Υπουργών στη συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας να περάσουμε σε μια πιο συστηματική προσέγγιση που είναι εξέλιξη στο πρώτο εξάμεινο του 2012 και μάλιστα αν επιβιώσουν οι Υπουργοί των ενδιαφέρον τους να πάμε και πιο πιο φιλόδοξες δράσεις όπως αυτές που υποστηρίζει η εξαιρετική έκθεση του κυρίου Λίζεκ με καινοτόμες προτάσεις δηλαδή που θα μας επιτρέψουν να πάμε πέρα από αυτά τα πρώτα συγκεκριμένα αποτελέσματα για μια πιο παγκόσμια, ε, πιο καθολική προσέγγιση και πιο φιλόδοξη προσέγγιση της συνένωσης και της κοινής χρήσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική διαφάνεια, ε, αυτό μας ενδιαφέρει. Επίσης, μας ενδιαφέρει να υπάρχει μεγαλύτερη σύγκληση ε, σχεδιασμού των ε, εθνικών αμυντικών σχεδίων και επίσης μας ενδιαφέρει να απτύξουμε τη μελλοντική γενιά δορυφόρων επικοινωνίας και την τεχνολογία υποπτίας και αναγνώρισης, παρακολούθησης και αναγνώρισης πληροφοριών επιτήρησης και αναγνώρισης. Τώρα, Φυσικά υπάρχουν ε, και θεσμικές δυσκολίες, είναι γνωστές ε, και εδώ ήθελα να επιμείνω. Και ε, καθώς κάθομαι και δίπλα από το στρατηγό Αντριάνο, θέλω να πω ότι παρά, πέρα, παρά το ότι υπάρχουν αυτές οι θεσμικές δυσκολίες, νομίζω ότι από κοινού κατορθώσαμε να κάνουμε μια πολύ σημαντική δουλειά, δηλαδή να δράσουμε έτσι ώστε να μην ε, υπάρχουν αντιπαλότητες μεταξύ των οργανισμών, αλλά δράσαμε και έτσι ώστε η αλληλοσυμπληρωματικότητα να είναι πραγματικότητα. Ε, κοιτάξτε, αυτό το απέτυχαν και τα κράτη-μέλη, το υπενθύμησαν και οι υπουργοί. Την ε, περασμένη εβδομάδα πολλοί υπουργοί είπαν ότι διαπιστώνουν ότι και από τις δύο πλευρές υπάρχει πραγματική συνεργασία που λειτουργεί. Έτσι λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, δεν ε, είμαστε μόνο εμείς ε, που το λέμε αυτό, το διαπίστωσαν και οι υπουργοί και μέσα από τις ε, εργασίες μας και μέσω από το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και κατορθώνουμε να παρουσιάσουμε για μια ακόμη φορά στα κράτη-μέλη μια υποστήριξη έτσι ώστε να μην υπάρχουν συγκρούσεις και να υπάρχει και συμπληρωματικότητα σε όσα κάνουμε. Κάτι άλλο που μου προκάλεσε εντύπωση, ε, πηγαίνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, υποστηρίζουν ε, ότι γίνεται, υποστηρίζουν ότι γίνεται στο ΝΑΤΟ, αλλά ότι γίνεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα. Μα είπαν ρητά ότι το υποστηρίζουν και μάλιστα συγκεκριμένα δήλωσαν την υποστήριξη αυτή ε, υπήρξε και δέσμευση συμμετοχή ορισμένε από τι συνεδριάσει του οργανισμού, στη συνεδρίαση που υλοποιούμε το Φεβρουάριο και ε, επίσης ε, θα ξεκινήσει και ένας διάλογος με ορισμένα από τα κράτη-μέλη μας, κυρίως για θέματα που αφορούν τη βιομηχανία και την αγορά. Τώρα, τα αποτελέσματα είναι σημαντικά. Προσπαθήσαμε να δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα ε, σε ό,τι αφορά τον τομέα κατανομή καθηκόντων. Ένα παράδειγμα είναι το εξή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες για τον αέριο ανεφοδιασμό. Ε, Έχουμε ε, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ που θα γίνουν οι εργασίες ε, για ε, τα αεροσκάφη παρακολούθηση στη θάλασσα περιπολία στη θάλασσα. Επίσης, όπως είπαμε, υποστηρίζουμε τον ιατρικό τομέα. Εμείς ε, υπό την ηγεσία της Ιταλίας αναπτύσσουμε κάτι τέτοιο, αλλά φυσικά βασιζόμαστε και στην τεχνογνωσία του ΝΑΤΟ, κυρίως ό,τι αφορά την τυποποίηση και βάση των διδαγμάτων του Αφγανιστάν. Τα ελικόπτερα αποτελούν ένα πολύ καλό παράδειγμα συμπληρωματικότητα. Ε, το ΝΑΤΟ ήθελε να ασχοληθεί με τι βιομηχανικέ πτυχέ ε, του εξοπλισμού και η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολήθηκε με τι πτυχέ τη κατάρτιση. Αυτό έγινε όπω γνωρίζετε έχουμε πάνω ε, από 120 πληρώματα ελικοπτέρων ε, που καταρτίστηκαν και τα μισά από αυτά χρησιμοποιήθηκαν στο Αφγανιστάν ε, υπό την πρωτοβουλία των κρατών μελών και μελών του ΝΑΤΟ στα πλαίσια του ΙΣΑΦ. Το ίδιο και για ε, τα εργαστήρια για την καταπολέμηση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και εκεί στα πλαίσια της ΙΣΑΦ ε, χρησιμοποιήθηκαν στο Αφγανιστάν ε, αυτές τις τεχνογνωσίες έτσι λοιπόν αυτή είναι η κοινή μας ε, δουλειά. Φυσικά αν είχε ρυθμιστεί και το θεσμικό πλαίσιο, αν, υπήρχαν, και αν υπήρχε το κατάλληλο πλαίσιο για την ανταλλαγή απόρριτων πληροφοριών, τότε αυτό θα ήταν ακόμη καλύτερο. Αλλά ε, βλέπετε τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματο. Και να κλείσω με το εξή. Δεν ε, υπάρχει θεωρικός περιορισμός που επιβάλλεται. Δηλαδή μια δράση όταν γίνεται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ή στο πλαίσιο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εμείς ε, υποστηρίζουμε τα κράτη στην απόφαση που θα λάβουν. Αυτό υπενθυμίστηκε από έναν υπουργό την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται λοιπόν για απόφαση των κρατών μελών. Εμείς απλώς παρέχουμε υποστήριξη και φυσικά μπορεί να υπάρξει ωφέλεια ε, από τα διάφορα θετικά που έχουν να προσφέρουν οι διάφοροι οργανισμοί. Έχουμε μια διατλαντική διάσταση μέσα από τον ΝΑΤΟ. Υπάρχει και μια διάσταση που σχετίζεται σε άλλες πτυχές πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Μιλάμε για την ε, συνέργεια με τις μη στρατιωτικές πτυχές και τη βιομηχανική διάσταση επί της οποίας ο Ευρωπαϊκός Οργανισμό Άμυνα έχει λάβει εντολή να εργαστεί.

Και μια παρατήρηση ακόμη για αυτές τις πτυχές συνέργειας με τις λοιπές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι κάτι που μας φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Για μας ε, είναι ένας ε, τομέας που θέλουμε να αναπτύξουμε συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φυσικά την ίδια στιγμή που υπάρχει οικονομική κρίση και την ίδια στιγμή που τα κράτη-μέλη πρέπει να αναπτύξουν αμυντικές ικανότητες, πολιτικές, ευρωπαϊκές πολιτικές ιδιαίτερα φιλόδοξες θα έχουν ένα αντίκτυπο και αρνητικό και θετικό στις πολιτικές άμυνας. Επίσης ε, έχουμε και το πρόγραμμα ΣΕΖΕΡ, ε, το πρόγραμμα του ενιαίου ουρανού, ε, που είναι ένα παράδειγμα και είχαμε προτείνει στο ΝΑΤΟ να προβεί σε μια διάρθρωση υπάρχει μια διάρθρωση έτσι ώστε οι ανάγκες ε, του ΝΑΤΟ και οι νόμιμες ενσυχίες του να λαμβάνονται υπόψη όταν ε, θεσπίστηκε ο νέος ουρανός και το ΣΕΖΑΡ. Έτσι λοιπόν γι' αυτό είχαμε μια ένα άτυπο φόρουμ και μπορούσαμε να κάνουμε την ίδια δουλειά σε ένα τομέα που παρακολουθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις ραδιοσυχνότητες, το ραδιοφάσμα και Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και τους εταίρους μας ε, στο ιστορικό της Επιτροπής να δημιουργηθούν όσο δυνατόν περισσότερες συνέργειες στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά υπογραμμίζεται και στην έκθεση της Επιτροπής σας. Και ένα ακόμη στοιχείο που έχει αναφερθεί επανειλημμένος είναι ένα στοιχείο βασικό για όλες τις προσπάθειες ανάπτυξης ε, αμυντικών ικανοτήτων, είναι ο συνδέσμος με τις πτυχές της αγοράς. Και λοιπόν ε, ταυτόχρονα ε, όσο υλοποιούμε αυτό το εγχείρημα μεταφέρουμε στο ιστορικό δίκαιο και το πακέτο της άμυνας και επίσης ε, την οδηγία περί δημόσιων προμηθειών στον τομέα της άμυνας ε, και εργαζόμαστε με την Κομισιόν, με τον κύριο Μπαρνιέ και έχουμε ε, και την Task Force ε, έτσι ώστε, που θα συστηθεί από τους κύριους Σταγιάννη και Μπαρνιέ έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ο καθένας ε, θα αναλάβει τις ευθύνες του έχει ευθύνη και η Κομισιόν για να γίνει σεβαστή συνθήκη και να θετηθεί σε εφαρμογή η οδηγία εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν με έναν κατάλληλο τρόπο ε, ε, το άρθρο της συνθήκης που έχει να κάνει με αυτό το τομέα της άμυνας. Λοιπόν, ε, αναφέρθηκα σε διάφορα στοιχεία, συνέργεια με τις άλλες πολιτικές της Ένωσης. Έτσι, λοιπόν, στα πλαίσιο αυτό έχουμε και τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και θεωρούμε ότι υπάρχει μια φυσική συμπληρωματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στρατηγέ, το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να λάβω το λόγο και πάλι ενώπιον τη Επιτροπή Ασφάλεια και Άμυνα και μάλιστα μετά την κυρία Αγνού. Θα ήθελα να πω ότι είναι εξαιρετικέ ε, οι αναμνήσεις μου από την περυσινή μου επίσκεψη και παρουσία στην Επιτροπή σας, που ήταν ε, μετά την ε, διάσκεψη της Θήκης τη Λισαβόνας και την εταιρική σχέση με το ΝΑΤΟ. Θα τηρήσω εξάλλου την εταιρική σχέση και στις γλώσσες που θα χρησιμοποιήσω για να υπάρξει κάποια ισορροπία. Τα δύο πρώτα χρόνια κατά τα οποία βρίσκομαι επικεφαλής ε, αυτής ε, της διοίκησης ε, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί. Προσπαθούμε να έχουμε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, με το Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη Μονάδα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρίσεων. Υπάρχουν ε, διάφορα ζητήματα όπως ε, η παγκόσμια προσέγγιση και αυτό το θέμα αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της Smart Defense, της έξυπνης ε, άμυνας που μου ανέθεσε ο κύριος Ράσμουσεν να προάγω και με την διάσκεψη που θα γίνει στο Σικάγο το Μάιο. Παράλληλα θέλουμε να έχουμε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη αυτού του στόχου και το πιο σημαντικό για να είναι πραγματικά βιώσιμη η πρωτοβουλία μας είναι να υπάρχει συνέργεια με αυτά τα οποία γίνονται στο ε, πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ανάλυση είναι μια ανάλυση με την οποία συμφωνούν τα διάφορα έθνη και έχω επισκεφθεί πάνω από 10 κράτη στα πλαίσια ε, ε, αυτής της προσπάθειας για την έξυπνη άμυνα και συνεχώς μου κάνει εντύπωση ότι ε, όλοι βρίσκουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με αυτή την πρωτοβουλία έξυπνης άμυνας. Θα ήθελα να σας παραθέσω τις δραστηριότητες της πρωτοβουλίας μας για την έξυπνη άμυνα πριν μιλήσω για τις σχέσεις που έχει αυτό με την προσπάθεια προσπάθεια συνένωσης και κοινή χρήση, το pooling and sharing σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν υπάρχει η διάσκεψη κορυφή τη Λισαβόνα, όπου ένα βασικό θέμα ήταν η επιθυμία μεταρρύθμισης, ξεκινώντας από την διάθρωση του οργανισμού και ε, περνώντας ε, σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη ικανοτήτων. Και μετά την Άνοιξη, όταν ε, είχαμε την οικονομική και δημοσιονομική κρίση, η οποία ήταν όλο και περισσότερο έντονη, ε, συνεχίστηκαν αυτές ε, οι συζητήσεις και την τωρινή κατάσταση δεν μπορούμε να δαπανούμε περισσότερα για την άμυνα. Σχεδόν όλες οι χώρες είναι έτοιμες και πρόθυμες να δαπανούν λιγότερα και πολύ λιγότερα. Άρα θα πρέπει να δαπανούν καλύτερα για να μην είμαστε ευάλωτοι από στρατηγικής πλευράς. Κατά την ορίμανση αυτή τη πρωτοβουλία όπου έπαιξε κεντρικό ρόλο η διαβούλευση με τον οργανισμό, υπάρχουν πολλοί άξονε και θα ήθελα να παραθέσω ορισμένου άξονες. Μία προσπάθεια ε, θέσης προτεραιοτήτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίως όταν μειώνονται οι πόροι. το, το ΝΑΤΟ μπορεί να έχει ένα τμήμα μόνο της ικανότητας της συμμαχίας ε, και όσο μειώνεται η συμμετοχή όλων, τόσο σημαντικότερη είναι η, τόσο σημαντικότερος είναι ο επιμερισμός. Χρειάζεται και ένας βαθμός εξειδίκευσης και παράλληλα συμφωνούμε με τις διεθνικές δράσεις. Έχουμε επισημάνει πολλές επιχειρήσεις που θεωρούμε βιώσιμες, περίπου 14 ε, είναι σε πολύ καλή εξέλιξη, ε, διότι προχωρούν συγκεκριμένες χώρες προς μια κατεύθυνση και αναλαμβάνουν δράσεις ε, σχηματίζοντας ομάδες χωρών με συνεκτική αντιμετώπιση. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται συνεκτικά, ακόμη και αν χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο ανάπτυξής τους. Αυτές είναι πρακτικές δράσεις της έξυπνης, έξυπνης άμυνας. Αυτό προωθείται εξάλλου και στο πλαίσιο του pooling and sharing στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίθεται το θέμα του αν αυτές οι πρωτοβουλίες ε, βρίσκονται ε, σε αντιπαράθεση και αν, ή αν είναι συμπληρωματικές. Νομίζω ότι έχουμε πλέον την απάντηση και η απάντηση είναι ενθαρρυντική. Ένας τρόπος να εξετάζουμε το θέμα είναι αν κάθε μία από τις πρωτοβουλίες μας θα ήταν καλύτερα να υπάρχει μόνη της χωρίς τις υπόλοιπες. Η δική μου άποψη είναι ότι αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοενισχύονται σαφώς. Πιστεύω ότι και οι δύο οργανώσεις και οι δύο οργανισμοί κάνουν παρόμοια διάγνωση και αυτό ενισχύει την αξιοπιστία των κρατών. Η βασική μας ανάλυση όσον αφορά τις μελλοντικές προκλήσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για να τις αντιμετωπίσουμε είναι παρόμοια η στρατηγική ε, έννοια ε, του ΝΑΤΟ και ε, η μακροπρόθεσμη αντίληψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας έχουν παρόμοιες απόψεις και έχουμε πάρει πολλά διδάγματα ημέν από τους δε. Σε, διάφορες, σε διάφορα παραδείγματα επιχειρησιακών δράσεων. Επίσης, σχέσεις ε, υπάρχουν ισχυρές άτυπες σχέσεις πριν από την έναρξη των πρωτοβουλειών και υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στα εγκαίνια πρωτοβουλειών όπως είναι ε, η ημέρα ε, για τον τομέα ε, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη βιομηχανία. Προσπαθούμε να έχουμε συγκεκριμένα παραδοτέα αποτελέσματα σε διάφορους τομείς όπως είναι τα αυτοσχέδια εκρηκτικά. Αυτή η σύγκληση μπορεί να δημιουργήσει μια διαφορετική ανησυχία. Μήπως τυχόν υπάρχει επικάλυψη στις ε, πρωτοβουλίες μας και αν υπάρχει επικάλυψη πώς μπορούμε ε, να την αποφύγουμε. Είναι ένα σημείο κέρια σημασίας και πιστεύω ότι η απάντηση εδώ είναι θετική, διότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολλές προσπάθειες εναρμόνισης. Στην πρόσφατη έκθεση του κυρίου Λίζεκ ε, ακριβώς αναφέρεται αυτό το θέμα και είναι πολύ ενθαρρυντικά αυτά που αναφέρονται. Σε θεσμικό επίπεδο βασιζόμαστε στην ε, καλή βούληση ε, και προσπαθούμε να υπάρχει αμοιβαία διαφάνεια και ανταλλαγή απόψεων και ανταλλαγή ιδεών, ιδίω μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα και τη δική μου διοίκηση. Έχω συναντηθεί με εμπειρογνώμονε και επιβεβαιώνω την προσπάθειά του. Ακριβώ λόγω αυτή τη αμοιβαία επίγνωση θα προχωρήσουν συμπληρωματικά σχέδια και η κυρία Αγνού πολύ σωστά ανέφερε το παράδειγμα των ελικοπτέρων. Άλλο ένα παράδειγμα είναι ότι και οι δύο έχουμε σχέδια για την ιατρική υποστήριξη και την, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διαρθρώνονται αυτά τα προγράμματα. Είναι απόλυτα συμβατά τα σχέδιά μας ε, και ε, αλληλοενισχύονται. Ε, η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρώνεται στο interface και η πλευρά του ΝΑΤΟ στις κοινέ προδιαγραφές. Και πέρα αυτών, πέραν των θεσμικών οργάνων, πιστεύω ότι τα σχέδια τα οποία προάγουμε θα αποτελέσουν ένα σημαντικό παράγοντα εξέλιξη αυτών των πρωτοβουλειών και τα κράτη-μέλη είναι αποφασισμένα να επιτύχουν και τα προγράμματα αυτά είναι ανοιχτά και στη συμμετοχή εταίρων εκτός ΝΑΤΟ, βέβαια κατόπιν πρωτοβουλίας των χωρών που έχουν την ηγετική πρωτοβουλία πρωτοβουλίες πολλαπλών κρατών συγκεντρώνουν χώρες ε, του ΝΑΤΟ και χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Και αυτό δεν είναι ένα βήμα στα τυφλά, είναι μια πραγματικότητα. Γνωρίζουμε ότι ε, υπάρχει συνεργασία όπως στην ε, περίπτωση του C-17. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η στρατηγική εγκύτητα μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών σε ένα πολυεθνικό πρόγραμμα. Και αυτή η εγκύτητα μπορεί να βασίζεται σε κριτήρια γεωγραφικά, πολιτιστικά, γλωσσικά, γεωπολιτικά, μια υφιστάμενη ιστορία συνεργασίας ε, και άλλα. Κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι ο στρατηγικό στόχο και των δύο πρωτοβουλειών είναι το να κρατήσουμε τι ικανότητε και των ε, δύο οργανισμών ε, χωρί να έχουμε περισσότερους πόρους, αλλά έχοντας μεγαλύτερη συνεργασία, μεγαλύτερη συνοχή, καθώ και καινοτομία την οποία να μπορούμε να πληρώσουμε. Εναρμονισμένη πρόσκληση και διαφρομένη χρήση των πόρων, τόσο ώστε να παραμείνουμε αξιόπιστοι και να, είμαστε, να έχουμε τη δυνατότητα να απαντούμε σε κρίσεις. Θέλουμε να ενισχύσουμε με τον ισχύοντα προϋπολογισμό την ικανότητά μας για αντιμετώπιση κρίσεων και ε, να δημιουργήσουμε ε, το δυναμισμό ε, στο πλαίσιο της έξυπνης άμυνας. Αυτό θα αυξήσει το δυναμισμό και για τη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δημιουργήσουμε μια πραγματική πρωτοβουλία για μεγαλύτερο συντονισμό και διαλειτουργικότητα. Αυτή η γόνιμη εμπειρία μπορεί να αποδείξει ότι όλοι μπορούν να βγουν κερδισμένοι από αυτή την ανοιχτή συνεργατική σχέση. Είναι ένα, δίδαγμα το οποίο θα μπορέσει να εφαρμοστεί και πολύ περαιτέρω από τα τωρινά μας προγράμματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, στρατηγέ. Ο κύριος Βανόρντεν θέλει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τους δύο προσκεκλημένους μας στο βήμα, την εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και τον εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που έρχεται η κυρία Αγνού στην Επιτροπή μας. Και πρέπει να σας πω που χαίρομαι πολύ το ότι που η Ιρλανδία θα αναλάβει την επιμόρφωση όσον αφορά τα ναυτικά θέματα. Είναι μια σημαντική ναυτική δύναμη. Δεν ήξερα ότι είχαν ναυτικό, αλλά μάλλον έχουν κάποιο ένα μικρό ναυτικό. Και βέβαια οι Ηνωμένε Πολιτείες επιθυμούν να υποστηρίξουν οτιδήποτε γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ουσιαστικά είναι απεγνωσμένοι για μεγαλύτερη συμμετοχή από τους Ευρωπαίους συμμάχους και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε επιτέλους να οδηγήσει σε έναν καλύτερο επιμερισμό του βάρους, του άχθους. Κάποια ερωτήματα θέλω να θέσω. Κύριε Στρατηγέ Αμπριάλ, μας μιλήσατε για τις διαφορές ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και το ΝΑΤΟ. Δεν είμαι όμως απόλυτα πεπισμένος. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι εσείς βρίσκεστε προτετελεσμένου γεγονότος και πρέπει να ασχοληθείτε με αυτό το τέχνασμα εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Θα ήταν πιο εύκολο να μην υπήρχε. Γιατί αν δείτε τις αμυντικές ικανότητες και σχετικές πρωτοβουλίες του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και όλες τις δραστηριότητες γενικότερα του ΝΑΤΟ, προφανώς όλες αυτές οι προτάσεις που ε, υποβάλλονται αυτή τη στιγμή είναι κοινέ για όλους τους στρατούς ουσιαστικά. Δεν υπάρχει κάποια κάποιο ιδιαίτερο ευρωπαϊκό χαρακτηριστικό ή κάποια ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα. Οτιδήποτε συζητάμε εδώ απασχολεί και το ΝΑΤΟ. Βοηθήστε με λοιπόν να καταλάβω ποια και πού βρίσκεται η προστιθέμενη αξία της περίφημης ευρωπαϊκής συμμετοχής και παρέμβασης, τη στιγμή που στα πλαίσια του ΝΑΤΟ μιλάμε για πάνω κάτω τις ίδιες χώρες. Μια εξαίρεση βέβαια θα είναι η Σουηδία που έχει πολύ σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις και ένα πολύ σημαντικό μια πολύ σημαντική αμυντική βιομηχανία, αλλά ακόμα βλέπω ότι και η Σουηδία ουσιαστικά συμμετέχει στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Επομένως βλέπω ότι σας πιέζουν, σας εξαναγκάζουν να προσαρμοστείτε κάπως την ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Απλώς δεν μπορώ να καταλάβω πού έγκυται η προστιθέμενη αξία. Με κάθε σεβασμό το λέω αυτό, κυρία Αρνού, ξέρω ότι και εσείς και οι συναδελφοί σας κάνετε μια εξαιρετική δουλειά. Όσον αφορά τώρα το pooling and sharing, πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτή η συνένωση πόρων τελικά θα είναι όντως διαθέσιμη όταν τη χρειαζόμαστε. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις στη Λιβύη, οι πρόσφατες επιχειρήσεις στη Λιβύη. Από ό,τι κατάλαβα, η Γερμανία αποσύρθηκε, απέσυρε τις δυνάμεις της από την στρατοτική μονάδα του ΝΑΤΟ που επέμβαινε στη Λιβύη και χρειάστηκαν να αντικαταστηθούν αυτές οι δυνάμεις της Γερμανίας. Κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο. Αναφέρομαι για τη μονάδα Άουαξ στη Λιβύη. Και στο παρελθόν υπήρξε ένα κράτος το οποίο ενώ κανονικά θα έπρεπε να δώσει κάποια πολεμοφόδια στα πλαίσια μιας κοινή αποστολής τελικά αρνήθηκε να παρέχει τα πολεμοφόδια αυτά σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της συμμαχίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτές τις δύσκολες στιγμές τελικά δοκιμάζεται και η πολιτική βούληση. Και τότε τελικά πολύ συχνά βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένε χώρες οι οποίες δεν έχουν μια σταθερή στάση για τα ζητήματα αυτά τα αμυντικά. Κύριε Στρατηγέ, αναφερθήκατε επίσης στην βελτίωση της ε, δύναμης ε, πολέμου ανάπτυξης. Είχαμε τους εκπροσώπους από την πρωτοβουλία της ε, Βαϊμάρης. Και από ό,τι φάνηκε, το τελευταίο πράγμα το οποίο σκέφτονται είναι η διεξαγωγή πολέμου ή διεξαγωγή μάχης. Από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να έχει δυνάμεις που μπορούν να σκοτώσουν ανθρώπους. Από ό,τι φαίνεται η δική μας ιδέα, η δική μας προσέγγιση είναι πολύ διαφορετική εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήμουν υπέρ της αύξησης των μαχητικών, των μάχημων μονάδων, αλλά από ό,τι βλέπω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινείται προς αυτό και όσον αφορά την αλληλοσυμπληρωματικότητα, την αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης και όσον αφορά την αξιοπιστία των συμμάχων στα πλαίσια του pooling and sharing. Θα ήθελα από αυτό να αναφερθείτε. Σας ευχαριστούμε κύριος Γιάννης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την κυρία για ε, τα συγχαρητήρια που έλαβε στο Συμβούλιο του 1η Δεκεμβρίου σε ό,τι αφορά την περιβόητη συνένωση και κοινή χρήση που λένε ξέρινγκ. Επίσης, ε, θέλω να συγχαρώ το στρατηγό Τριάλ, ο οποίος ε, παρευρέθη σε αυτή την επιτροπή πριν ένα χρόνο. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί ε, μπορώ να σας πω ότι εμείς, πάρα πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Βουλίου, είμαστε σύμφωνοι στο εξή, στο να υπάρχει μια σταδιακή πολιτική για να σημειώσουμε πρόοδο στην οικονομήση μιας ε, κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας στην Ευρώπη. Ενίοτε έχω την εντύπωση στις συζητήσει αυτές της Επιτροπής ότι το θέμα Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ, τουλάχιστον για ε, συναδέλφους, ε, σε ορισμένους συναδέλφους, φαίνεται να τους ξυπνά κάτι που να μοιάζει περισσότερο με αυτές ε, τις ε, θεολογικές συζητήσεις ε, που υπήρχαν στο Μεσαίωνα από ότι και αφορά το ποιος είναι ο ρόλος του καθένα στην πράξη. Εγώ δεν είμαι τόσο μπερδεμένο ε, σε σχέση με αυτά τα θέματα. Εγώ ε, θεωρώ ότι εδώ μιλάμε για συμπληρωματικούς ε, στόχους και για συμπληρωματικές λειτουργίες που βασίζονται σε κοινέ αξίε. Έτσι λοιπόν ε, δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερο ΝΑΤΟ σκεφτόμενοι ότι αυτό μποϊκοτάρει την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκή ε, κοινή Ασφάλεια και άμυνα, ή να λέμε ότι αν έχουμε καλύτερη ευρωπαϊκή διάσταση αποδυναμώνεται το ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι και τα δύο οδεύουν προς την ίδια κατεύθυνση. Ε, μιλήσαμε για λευσιβληματικότητα, για μη επικαλύψει αναζήτηση ε, συνεργασίας, ε, βελτιστοποίηση. Μιλήσαμε και για την πρωτοβουλία της Βαϊμάρης, μιλήσαμε για την ευέλτιστη χρήση των πόρων. Όταν ε, έχουμε οικονομικές δυσκολίες, και το υπενθύμησε ο πρέσβης τη Ισπανίας μας είπε ότι ε, οι προϋπολογισμοί ε, και των 27 ε, ξεπερνούν τα 2 δις. Αλλά το θέμα είναι ότι δυστυχώς δεν, δεν έχουμε ένα κοινό προϋπολογισμό. Πάντως, στο μέτρο του δυνατού θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους αυτούς. Εγώ προσωπικά και λέω εγώ, δεν μιλώ εξ ονόματος της χώρας μου. Ξέρετε ότι εμείς εδώ τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τοποθετούμαστε και λέμε και την προσωπική μας άποψη. Ε, έτσι λοιπόν, ούτε εγώ εκπροσωπώ την ομάδα μου, όμως μπορώ να σας πω ότι είμαι ε, κάπως πιο διστακτικός ε, απέναντι σε αυτό που ιστορικά αναφέρεται ότι το ΝΑΤΟ εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν οι Ηνωμένες ε, θέλουν εμείς να ε, είμαστε όλο ένα πιο υπεύθυνοι, όλο ένα πιο ανεξάρτητοι. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να είμαστε κι εμεί όλο ένα ε, πιο υπεύθυνοι για τη δική μας ε, πολιτική. Ε, είχαμε και τον ε, πόλεμο στο Ιράκ ε, και ξέρετε τις Ηνωμένες Πολιτείες τότε δεν τις ανδιέφερε αυτή η αυτόνομη δυνατότητα σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια της Ευρώπης 60-70 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πρέπει όλο ένα και περισσότερο εμείς να υλοποιούμε τη δική μας άμυνα. Είναι δική μας ευθύνη αυτό. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την παρουσία σας εδώ. Εμένα πραγματικά με διαφωτίσατε. Merci. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σαγκουράκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχήν θα συμφωνήσω με την επισήμανση του στρατηγού κυρίου Αμπριάλ ότι ενδεχομένως στις περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει μείωση των στρατιωτικών δαπανών. Δυστυχώς αυτό δεν αφορά την Ελλάδα, τουλάχιστον όσον αφορά το πρόγραμμα των εξοπλισμών και το πρόγραμμα των ατοικών υποχρεώσεων. Για τα μεν εξοπλιστικά προγράμματα η χώρα μου θα δαπανίσει το 12-22% παραπάνω από το 11% και για τα ανατοϊκά ε, εξοπλιστικά προγράμματα 60%. Άρα σωστό είναι αυτό ότι δεν αφορά όλους. Όμως ε, θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση στον ε, στρατηγό μας ούτως ή άλλως είτε μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση είτε μιλάμε για ΝΑΤΟ, μιλάμε για επιχειρήσεις εκτός ορίων. Όλα τα προγράμματα τα οποία συζητάμε είναι επιθετικά προγράμματα. Κανένα δεν έχει να κάνει με την έννοια της, ε, ε, εδαφικής, της υπεράσπισης της εδαφικής ακαιρεότητας των χωρών μελών, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του ΝΑΤΟ. Γιατί εγώ να μην πιστεύω και να μην λέω ότι το ΝΑΤΟ και με βάση τη στρατηγική της Λισαβόνας και με βάση τα όσα υπόθηκαν και με βάση την έξυπνη, τα έξυπνα εξοπλιστικά προγράμματα ετοιμάζεται για όλο και πιο μεγάλες, όλο και πιο μαζικές, όλο και πιο φωνικές θα πω επιχειρήσεις σε κάθε σημείο της γης. Αν αυτό είναι γεγονός, τότε ρωτάω γιατί δεν μειώνονται τουλάχιστον οι εξοπλισμοί εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την εδαφική άμυνα των χωρών μελών. ή άλλως επιθετική είναι η πόλεμη που γίνονται. Όλοι αυτοί. Τα τελευταία 20 χρόνια αυτό γίνεται. Γιατί, γιατί αυτό το διπλό παιχνίδι. Και όσον αφορά την κυρία Αρνού, θα ήθελα να την παρακαλέσω, αν κατάλαβα καλά από την τοποθέτησή της, μίλησε για ορισμένες στριβές, ορισμένες ε, διαφοροποιήσεις μεταξύ θεσμών. Μπορεί να μην άκουσα καλά, μπορεί να είναι θέμα μετάφρασης. Ε, αν είναι έτσι, σε τι αναφέρεται. Και τέλος, θα ήθελα μια διόρθωση. Επειδή άκουσα δύο φορές να λέγεται ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2,5 δις ευρώ, είναι λάθος. Με βάση τη μελέτη που έχουμε διαβάσει για το ε, pooling and sharing, είναι 200 δις ευρώ το χρόνο οι αμυντικές δαπάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 700 δι στι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι 2,5 δι όπως ακούστηκε. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Αρνού για την uh, πολύ καλή παρουσίαση που, κάναμε, που έκανε εδώ πέρα, καθώς επίσης και για την φιλοξενία της στα πλαίσια του, της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας είναι η κυρία Άστον. Πόσο συχνά έρχεται στην έδρα σας. Πόσο συχνά ήρθε κατά τη διάρκεια της θητείας της. Πρώτο ερώτημα αυτό. από ό,τι έχω μάθει δεν σας έχει επισκεφθεί ακόμα και αυτό με ανησυχεί, αλλά θα ήθελα να μου το διευκρινίσετε εσείς. Δεύτερον, είπατε ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Ποιο πιστεύετε όμω ότι είναι ο τελικός προορισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα, Εσεί εργαστήκατε για το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, κάνατε μια καταπληκτική σταδιοδρομία και δεν ξέρω αν προσπαθήσει να κάνετε αυτό που απέτυχε να κάνει ο Σούμαν το 1954 όταν ήταν υπουργό εξωτερικών, δηλαδή να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή κοινότητα Άμυνα. Αυτό είναι ο απότερο στόχο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα. Ευχαριστώ και πριν δώσω το λόγο πάλι στην κυρία Γνού και στον στρατηγό Αβδιάλη, θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με τα υλικά και τις έρευνες για, ε, τον εξοπλισμό, για τους εξοπλισμούς, ε, πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι οργανισμοί δεν, δεν κάνουν έρευνα για υλικά τα οποία απευθύνονται σε επιθετική χρήση. Υπάρχουν στρατιώτες κάποιων κρατών μελών που υπηρετούν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, το τονίζω αυτό, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν παραδείγματο χάρη και κάποιοι από αυτούς έχουν και σκοτωθεί. Η δουλειά που έχει γίνει από τον οργανισμό για την ιατρική υποστήριξη ή για τα εργαστήρια κατά των ε, αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Όλη αυτή η ερευνητική δουλειά είναι δουλειά ε, για την προστασία των πολιτών. Ε, οι στρατιώτες μας υπηρετούν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και επομένως υπό την μεγαλύτερη διεθνή νομιμότητα. Ας έχουμε λοιπόν τον ε, δέοντα σεβασμό προς τους στρατιώτες αυτούς, προς τις οικογένειες αυτών των στρατιωτών που πέφτουν θύματα ε, αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και γι' αυτό ήθελα να κάνω αυτή τη διευκρίνηση τώρα. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Αγνού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάντοτε είναι χαρά μου να προσπαθώ να απαντώ στον κύριο Βανόρντεν. Λέτε ότι συνεχίζετε να, να δυσκολεύεστε, να καταλάβετε πώς μπορεί ο στρατηγός Αμπριάλ ε, να συνδυάσει αυτά τα οποία κάνει με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. πρέπει να δούμε αν πραγματικά μιλάμε σοβαρά για την συνέργεια, για μεγαλύτερες ικανότητες, ε, γιατί αν όντως μιλάμε σοβαρά και αν όντως βλέπουμε κατάματα την πραγματικότητα, τη σημερινή πραγματικότητα, δεν θα έπρεπε να παραμελούμε τη συνεισφορά της Ιρλανδίας. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να έχουμε μεγαλύτερες ικανότητες. Όλοι μαζί όμως. Δεν λέμε ότι η μία ή οι δύο χώρε μπορεί να κάνουν κάτι περισσότερο. Ξέρουμε ότι κάποια κράτη-μέλη είναι μεγαλύτερα όσον αφορά την άμυνα και καλά κάνουν. Αλλά ένα από τα πράγματα ε, ε, τα οποία περιλαμβάνονται στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και είναι και κάτι που το κάνουν και οι Αμερικανοί. Δεν λέμε συστηματικά ότι επειδή το κάνουν οι Αμερικανοί θα πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Αλλά παρόλα αυτά, ε, ας είμαστε ρεαλιστές θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω οι Ευρωπαίοι συλλογικά. Στην προηγούμενη θέση μου είχα δει ότι η Ιρλανδία συμμετείχε στην επιχείρηση στο Τσάντ και ανέλαβε σημαντικές ευθύνες και πιστεύω ότι ήταν θετικό αυτό για την ευρωπαϊκή δράση. Η Ιρλανδία νησί είναι, έχει σχέση με τα ναυτικά θέματα. Όταν βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι έχει ε, ευθύνη για εκπαίδευση στον τομέα του ναυτικού και υπάρχει και εδώ κάποια εξέλιξη, όπως είπε και ο Υπουργός της, για τα θέματα της δράσης. Ε, πιστεύω ότι είναι θετικά αυτά. Πάντοτε βέβαια στο πλαίσιο του ΟΗΕ που συζητάμε, είναι ένα θετικό στοιχείο. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στον τομέα των ικανοτήτων, είναι όχι μόνο να αυξάνουμε τις ικανότητες των κρατών μελών που έχουν τη μεγαλύτερη ικανότητα αυτή τη στιγμή, αλλά να αυξάνουμε τις ικανότητες που θα παίξουν το ρόλο καταλήτη για την κοινή μας δράση. Και τονίζω ότι για μένα είναι σημαντικό το ότι μια χώρα σαν την Ιρλανδία μπορεί τώρα να υποστηρίξει μεγαλύτερες ικανότητες και είναι έτοιμη να παίξει ένα πραγματικά ενεργό ρόλο. Επίσης, αν αντιμετωπίζουμε με σοβαρό τρόπο τις συνέργειες και τη συνεκτική προσέγγιση, οτιδήποτε κάνουμε ε, τα στρατιωτικά, εμείς στρατιωτικά μέσα που χρησιμοποιούμε, τις τεχνολογίες, ε, τις τεχνολογίες ε, γεφύρωσης, είναι πολύ σημαντικά και θέλουμε να δουλέψουμε μαζί με την Επιτροπή για το καινούριο ΙΕΣ, για το διάστημα, για την ε, παρακολούθηση στη θάλασσα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στον τομέα των συνεργειών. Και αν δείτε την πραγματικότητα σήμερα, δεν θα σας εκπλήξει το ότι ο στρατηγός Αμπριάλ θα δεχτεί να λάβει υπόψη του και να συνεργαστεί με την, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Τώρα για τη δεύτερη παρατήρησή σας για το θέμα της αξιοπιστίας των ικανοτήτων μας. Αυτό είναι ένα σημείο κλειδί και συμφωνώ απολύτως μαζί σας επ' αυτού. είναι κάτι στο οποίο καταβάλουμε προσπάθειες και είναι ένα ζήτημα και για τον στρατηγό Αμπριάλ και για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και για οποιαδήποτε διμερή συνεργασία αποτελεί ζήτημα. Και είναι ένα ζήτημα που έχει βρει κάποια λύση στο θέμα της διμερούς συνεργασίας όπως είναι η Γάλλο-Βρετανική στο πλαίσιο της ΝΟΤΕΦΚΟ και συμφωνώ με αυτό το είπε ο στρατηγό Αβριάλ για κάποια συμπλέγματα συνεργειών. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο στοιχεία ω απάντηση στην ερώτησή σα. Ένα στοιχείο είναι ε, ε, πολιτισμικό πολιτικό, στρατηγικό, κοινά πολιτισμικά στρατηγικά στοιχεία και το άλλο στοιχείο είναι κάποια πιο νομικά ζητήματα, κάποιες ρήτρε που μπορούν να βρεθούν, κάποια βρεθήκαν, βρέθηκαν κατά την επιχείρηση στη Λιβύη όσον αφορά την αερομεταφορά και νομίζω ότι και στα δύο σημεία αυτά πρέπει να δουλέψουμε. Και αν έχουμε επιμερισμένη χρήση, αν έχουμε κοινή στρατηγική άποψη, πιστεύω ότι μπορούμε να ωφεληθούμε και μπορούμε να βασιστούμε σε ρήτρε που δούλεψαν σωστά και να κάνουμε ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, γιατί πιστεύω ότι αυτά είναι εξαιρετική σημασία και συμφωνώ απολύτως μαζί σας αυτό που είπατε. Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή σας, ε, κύριε Γιάννη. Πιστεύω ότι η σχέση μας με τις Ηνωμένε Πολιτείε. είναι θετικό το ότι λέμε ότι δεν πρέπει να εξαρτώμεθα συστηματικά από τους άλλους. Είναι ε, για μας ένα καμπανάκι και Στις Ηνωμένε Πολιτείε μας λένε ότι έχουν κάνει τις μεγαλύτερες περικοπές στον τομέα της άμυνας, τις μεγαλύτερες περικοπές του προϋπολογισμού, δεν ξέρω αν είναι οι μεγαλύτερες ε, ε, ιστορικά ή μόνο οι μεγαλύτερες τον τελευταίο καιρό. Πάντως το θέμα της αλληλεγγύης είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, όχι γιατί δεν το θέλουν, αλλά γιατί μπορεί λόγω των περικοπών να μην είναι σε θέση να το κάνουν. Δεν θα προσθέσω τίποτα σε αυτά που είπε ο κύριος πρόεδρος, ο Ανόνταν Ζων, για το ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουμε δεν είναι επιθετικές και τα παραδείγματα ε, που δόθηκαν είναι πολύ καλά. Η ιατρική υποστήριξη, παραδείγματο χάρη. Όταν μιλάμε όμως ε, για πυρομαχικά, για ε, πυρομαχικά ακριβία και για αναγνώριση ακριβίας, θα πρέπει να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Και η μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγουμε θύματα, θύματα και δικών μας στρατιωτών, και για να ελαχιστοποιήσουμε τις παράπλευρες ζημίες για τους ε, επιτόπου πληθυσμούς. Και τα όπλα, που είναι όπλα ακριβίας, είναι απολύτως απαραίτητα όταν πρέπει να διεξαχθούν κάποιες ανθρωπιστικές αποστολές στο πλαίσιο μιας ανθρωπιστικής αποστολής. Και είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι και αυτές οι ικανότητες είναι δεοντολογικά και νομικά απαραίτητες εάν θέλουμε να δράσουμε. Και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ομόφωνη συμφωνία για ανθρωπιστική δράση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Κύριε Κάμπελ, ε, δεν θεωρείται επίσκεψη ε, επίσκεψη από την Βαρόνια γιατί είναι δικό τη οργανισμό. Σε σπίτι τη βρίσκεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα. Αυτό λέω ω απάντηση προ εσά. Τι είναι απόλυτε πληροφορίε το αν έχει έρθει ή όχι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι συνεργασίας και νομίζω ότι συνεργάζεται μαζί μας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας συνεχώς η Βαρονιά Τώρα για το ποιος είναι ο στόχος που ρωτήσατε. Νομίζω ότι ο στόχος είναι να υποστηρίξουμε αυτό το οποίο είναι έτοιμα να κάνουν τα κράτη-μέλη. Είναι κυρίαρχες οι αποφάσεις που λαμβάνουν στον τομέα των ικανοτήτων, παραδείγματο χάρη. Εμείς ως Ευρωπαϊκός Οργανισμό Άμυνα, είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη να λάβουν κυρίαρχε αποφάσει όσον αφορά την ικανότητα άμυνας. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη θέλουν να είναι αποτελεσματικά σε σχέση με το κόστος και να υπάρχει και διαλειτουργικότητα. Όλα τα θέματα που συζητάμε με τους υπουργούς αποσκοπούν στο να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί, να έχουμε καλύτερες ικανότητες στην Ευρώπη και ένα από τα κλειδιά για την καλύτερη ικανότητα είναι το να μπορούμε να συνεργαζόμεθα και να υπάρχει αποτελεσματική διαλειτουργικότητα. Αυτός είναι ο στόχος προς το παρόν. Τα υπόλοιπα θα είναι πολιτικέ αποφάσει που θα πρέπει να ληφθούν από τα κράτη-μέλη στη υψηλότερο επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι καθώ ε, κύριε μου, μίλησε ε, ε, μπορώ να μιλήσω κι εγώ γαλλικά αφού μίλησα αγγλικά να σας πω τώρα 21 και 44 21 είναι ο αριθμός αριθμών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και έχουμε 13 χωρίς διαφορά που δεν ανήκουν παρά στον ένα ε, οργανισμό και από τις δύο πλευρές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ΝΑΤΟ και πρέπει εμείς ε, νομίζω ότι ε, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν έχουν οι δύο οργανισμοί ούτε τα ίδια οράματα ούτε τους ίδιους στόχους και επίσης ακόμη και για τα ίδια θέματα μπορεί να πρέπει ε, να υπάρχουν και κάποιοι διαφορετικοί στόχοι. Ε, Πολλέ φορέ όμω εμεί ε, συνεργαζόμαστε για διάφορα θέματα και τελικά τα καταφέρνουμε για να αποφύγουμε τι επικαλύψει και να καταλήξουμε στο να έχουμε συμπληρωματικότητα στα σχέδιά μα. Και όταν λέω συμπληρωματικά να είναι τα σχέδιά μα, δηλαδή δεν ικανοποιούμαστε μόνο από το ότι θέλουμε να κάνουμε δύο φορέ τέτοια πράγματα αλλά αναλαμβάνουμε ένα πρόβλημα και μπορεί να βλέπουμε τις διάφορες πτυχές του και να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό στις διάφορες πτυχές του ή σε διάφορα στάδια, παραδείγματος χάρη. Νομίζω ότι ο κατάλογος ε, των ε, εργασιών μας ε, σας δείχνει ότι είναι προφανή τα πράγματα και εμείς από τη δική μας πλευρά ήδη έχουμε project που έχουμε εντοπίσει και στα οποία θα συμμετάσχουν και έθνη που ανήκουν μόνο στο ΝΑΤΟ και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω ότι το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει και από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία στο να συνεργαστούμε και οι δύο σε ένα παγκόσμιο επίπεδο για να υπερασπίσουμε παγκοσμίω την ασφάλεια και την άμυνα. Το ότι αφορά τώρα την εγγύηση των ικανοτήτων ε, και τη διάθεση των ικανοτήτων είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και είναι ένα θέμα στο οποίο συζητώ σε κάθε πρωτεύουσα που επισκέπτομαι για το Smart Defense, για αυτή την ευφυή άμυνα, είναι πραγματικά απαραίτητο, επιτακτικό, κάθε έθνος μεμονωμένα να λάβει υπόψη την έννοια της ισορροπίας μεταξύ της ελληνικής και της εθνικής κυριαρχίας. Κάθε απόφαση συμμετοχής ε, σε ένα project ε, λαμβάνεται φυσικά ε, ανεξάρτητα και φυσικά όταν έρθει κατάλληλη μέρα το κράτος θα αποφασίσει αν θα θέσει στην ε, διάθεση του οργανισμού ε, αυτές τις ικανότητες. Δεν υπάρχει μία και μόνη απάντηση, εξαρτάται από την πολιτική διαδικασία, από την κουλτούρα του καθέθνους, είναι ένα δύσκολο θέμα, αλλά φυσικά πρέπει αυτά τα θέματα να τίθονται ανάντι. Όταν ε, μιλώ για fighting power, Ξέρετε, γνωρίζετε τα άρθρα 4 και 5 ε, της Ουάσιγκτον που αναφέρει ε, ποιες θα μπορούσαν να είναι οι αποστολές μας. Φυσικά το ΝΑΤΟ έχει ένα επίπεδο φιλοδοξίας που είναι σαφώς προσδιορισμένο και μπορώ να σας πω ότι και στην ε, τελευταία μας εντολή ήταν η επιχείρηση στη Λιβύη και για να αντιμετωπίσουμε και να σεβαστούμε αυτό το σύνολο των κριτηρίων πρέπει να έχουμε ικανότητες που να μας επιτρέπουν ε, να αναπτύσσουμε ε, τις επιχειρήσεις μας σε όλα τα πιθανά φάσματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτό το fighting power, αυτές τις μάχημες ε, ικανότητες ε, και νομίζω ότι αυτό αφορά και τα έθνη που αποτελούν τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τώρα τον τρόπο που εργαζόμαστε. Εργαζόμαστε με μικρά βήματα. Εμεί προσπαθούμε να σεβόμαστε φυσικά το πολιτικό πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο θεσμών, αυτή η πολιτική μικρών βημάτων ή μιας ε, λογικής προσέγγιση, ε, φαίνεται επίση και από το ίδιο το οικοδόμημα του Smart Defense, δηλαδή αυτή τη ευφυού ε, Άμυνα, Προσπαθούμε να ε, διαλέξουν ε, τα ίδια τα κράτη ποια ομάδα θα σχηματίσουν ε, για να αναλάβουν το τάδε project και αυτό το σύνολο των ομάδων μας επιτρέπει να περάσουμε στο ανώτερο επίπεδο δηλαδή να έχουμε μια καθολική συνέπεια και συνάφεια και ε, στη δική μου περίπτωση το ΝΑΤΟ ε, θα έχει τις απαραίτητες ικανότητες για να αντιμετωπίσει τις φιλοδοξίες που ανέφερα προηγμένως. Και όπως ε, είπε και η Γενερούς στις εργασίες αυτές, κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι η αμοιβή εμπιστοσύνη. Και μπορώ να σας πω ότι οικοδομείται αυτή η αμοιβή εμπιστοσύνη, δεν μπορεί να προκύψει διαφορετικά. Και θα έλεγα ότι οι συνθήκες δεν είναι ίσως ιδανικές, αλλά πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου να μπορούν τα κράτη να διαλέξουν με ποιον θα εργαστούν. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο φετηρία. Τώρα, η εξαρτήσή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να επαναλάβω σε είπε συνάδελφος. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους Ευρωπαίους και είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό για τους Αμερικανούς και θα πρέπει και οι ευρωπαϊκές χώρες να συνειδητοποιούν αυτή την αλληλεξάρτηση και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σε ό,τι αφορά τώρα τη φύση των ε, σχεδίων επί των οποίων εργαζόμαστε, ε, φυσικά και εγώ δεν συμφωνώ με τον όρο που χρησιμοποιήθηκε επίθεση, αλλά ε, θα ήθελα να σας πω ότι ε, όταν ε, βλέπω ότι εργαζόμαστε για την υλικοτεχνική υποδομή, παραδείγματο χάρη οχήματα που μπορούν ε, να αντισταθούν σε κάποιε επιθέσει, σε κάποιε ενέδρε ε, και στι νάρκε, ε, μπορώ να σας πω ότι εδώ, παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα κλασικό σενάριο άμυνα και στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ελικόπτερα Όταν εργαζόμαστε για την κατάρτιση των πιλότων, το ίδιο ισχύει. Όταν ε, εργαζόμαστε επί των ε, αεροσκαφών για τις θαλάσσιες περιπολίες, μπορώ να σας πω ότι εκεί λαμβάνουμε υπόψη τη συλλογική άμυνα για να περισπίσουμε τις φιλοπικοινωνίες, παραδείγματος χάρη όταν ένα κράτος μέλος ε, μας πρότεινε ε, πρόσβαση των γυναικών ε, σε, κάποια, σε κάποιες θέσεις αμυντικές, δεν νομίζω ότι εκεί μιλάμε για επίθεση και έτσι λοιπόν ε, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτά τα project περιορίζονται σε ένα είδος επιχείρησης και όταν λέτε, επειδή εγώ θα έλεγα μάλλον ανάπτυξη, εξωτερικές επιχειρήσεις, ε, δείτε τη γεωγραφία. Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί για τη συλλογική άμυνα στο εσωτερικό της συμμαχίας και αν ε, πρέπει, παραδείγματος χάρη, ε, μια χώρα στον Νότο να συνεισφέρει ε, για να ωφελήσει μια χώρα του Βορρά. Ε, μπορώ να σας πω ότι έχουμε μια εσωτερική επιχείρηση ανάπτυξης και στη συνέχεια αν τα κράτη-μέλη, τα έθνη μέλη αποφασίσουν συλλογικά να συμμετέχουν σε μια εξωτερική επιχείρηση, τότε δεν βλέπουμε να υπάρχει αντίθεση στην ικανότητα ανάπτυξη και του ότι αυτές οι ικανότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογική άμυνα, στο πλαίσιο συλλογική άμυνας. Αυτά, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, στρατηγέ. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο, θεωρώ τα πάντα ήταν ε, σαφέστατα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις διευκρινήσεις σας, ε, κύριε στρατηγέ. Θα ήθελα να σας ζητήσω να περάσετε πάλι να μας δείτε μετά την σύνοδο του Σικάγο οι προηγούμενοι σύνοδοι του ΝΑΤΟ ήταν ε, σίγουρα μάλλον πιο εύκολες ε, για σας ε, να έρθετε να μας δείτε μετά τη Λισαβόνα για παράδειγμα, αλλά ελπίζω ότι και μετά το Σικάγο θα μπορέσετε να έρθετε να μας δείτε για να με ενημερώσετε. Κυρία Αρνού, εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, γνωρίζουμε πού βρίσκεται ο οργανισμός σας, επομένως θα χαρούμε πολύ να σας ξαναδούμε, να έρθουμε εμείς να σας δούμε Είδαμε ποια, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες του οργανισμού σας και ανεξάρτητα από τις πολιτικές παρεμβάσεις που θα γίνουν από την ύπατη εκπρόσωπο και την, την οποία θα ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, πιστεύω ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να βλέπουμε και εσά προσωπικά για να μας ενημερώνετε για την διαδικασία επίτευξης των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Εδώ και δύο χρόνια μιλάμε πολύ για την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνα και για την χρησιμότητα και το ρόλο που μπορεί να διεξάγει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Ακούστηκαν πολλές αμφιβολίες και υπήρχαν διάφορα ερωτηματικά στην αρχή. Θεωρώ όμως ότι κινούμαστε στο σωστό δρόμο. Υπήρξε, υφίσταται ακόμα μια διαδικασία εξορθολογισμού και μας εξήγησετε κι εσείς ότι υπάρχουν κάποια απτά πλέον πρακτικά σχέδια τα οποία εφαρμόζονται τα οποία είναι πολύ σημαντικά πέρα από την στρατηγική πτυχή την οποία τη γνωρίζουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η έμπρακτη εφαρμογή των σχεδίων του οργανισμού σας θα μας βοηθήσει να καταφέρουμε να ελοποιήσουμε κάποια προγράμματα συνένωσης και επιμερισμού. Πρόκειται για κάποια μικρά βήματα που γίνονται αυτή τη στιγμή που θα έχουν όμως πολύ σημαντικές συνέπειες. Είμαστε υπόλογοι και απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι είναι και Ευρωπαίοι φορολογούμενοι είναι πολύ σημαντικό να καταφέρνουμε και εμείς στη δική μας τη θέση να δείχνουμε προς τα έξω προς τους πολίτες μας ποια είναι η πρόοδος η οποία επιτυγχάνεται και σε ποιους τομείς δραστηριοποιούμεθα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη θεσιμότητά σας, για την παρουσία σας εδώ σήμερα και θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί προκειμένου να ενημερωθούμε ακόμα περισσότερο για τους τομείς δραστηριότητάς σας. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα δύο λεπτών, προτού προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που έχει να κάνει με την ομάδα COARM. Euh, Για το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πασκού θα αναλάβει την Προεδρία. Ευχαριστώ.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 Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω τον κύριο Φάμπιο Ντελαπιάτσα, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΚΟΑΡΜΑ, της Ομάδας Εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Όπλα, και μαζί του θα συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα τον ε, έλεγχο των εξαγωγών ε, στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού. Ζήτημα το οποίο μας ε, απασχολεί όλους, μας ενδιαφέρει όλους και ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται στην καρδιά πολλών άλλων συζητήσεων. Νομίζω ότι υπάρχουν διάφοροι καονισμοί που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το ζήτημα. Έχουμε οκτώ κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούνται και είμαι σίγουρο ότι η συμβολή του συναδέλφου μας θα δώσει έναυσμα για μια συζήτηση που θα ακολουθήσει. Κύριε Ντελαπιάτς, έχετε το λόγο. Uh, ευχαριστώ κύριε Πάσκου και καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Προκειμένου να ενημερώσω την Επιτροπή σας για τις δραστηριότητες της ΚΟΑΡΜΑ ε, κατά τη διάρκεια του 2011. Όπως θα γνωρίζετε, η ύπατη εκπρόσωπος με διόρισε ε, μόνιμο επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εξοργίες Συμβατικών Όπλων, ΚΟΑΡΜΑ. 1η Ιανουαρίου ανέλαβα τα νέα μου καθήκοντα, επομένως περίπου ένα χρόνο εργάζομαι για το αντικείμενο αυτό. Σήμερα είναι η πρώτη μου ευκαιρία να συνεχίσω την παράδοση αυτή που ξεκίνησε το 2004 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή να προβλέπετε μία ακρόαση, μία δυνατότητα ακρόασης με τον πρόεδρο της ΚΟΑΡΜΑ. Το 2009 ήταν η τελευταία τέτοια ευκαιρία κατά τη διάρκεια της Ιουδική Προεδρίας και κατά τη διάρκεια του 2010, καθώς επίσης και το πρώτο εξάμεινο του 2011, δεν κατέστη δυνατό να διοργανωθεί τέτοια ακρόαση λόγω διαφόρων αιτιών όπως το ότι ε, δημιουργούσαμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής δράση, έπρεπε να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα και άλλαξε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισηγητή για τα ζητήματα αυτά. Επομένω, ε, θα ήθελα να επικεντρωθούμε σήμερα στην παρουσίασή μου, σε μια σύντομη ουσιαστικά παρουσίαση, προκειμένου να ακούσω και τι δικέ σα ερωτήσει, Να επικεντρωθώ λοιπόν στι δραστηριότητε ε, που βρίσκονται στις προτεραιότητες της ΚΟΑΡΜΑ και να δούμε και πού θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας κατά τη διάρκεια του 2012. Επίσης, ελπίζω ότι τους επόμενους μήνες θα μας σε θέση να, αναστήσουμε, να, να την παράδοση αυτή της εξάμηνης ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την ΚΟΑΡΜΑ και ελπίζω και εγώ και οι συναδελφοί μου στα πλαίσια της ΚΟΑΡΜ να είμαστε σε θέση να σας ενημερώνουμε για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο Συμβούλιο για ζητήματα άμυνας και εξαγωγών όπλων. Και κατά αυτόν τον τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επιτελέσει και το έργο του, α, της επιτήρησης δηλαδή των αποφάσεων που λαμβάνονται στο Συμβούλιο. Καταρχάς, να σας δώσω κάποιες ε, λεπτομέρειες ε, όσον αφορά την ε, εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ΚΟΑΡΜΑ. Βασικός μας στόχος είναι να εξασφαλίσουμε ότι εφαρμόζεται η κοινή θέση του Συμβουλίου 944 του 2008, μια κοινή θέση λοιπόν του Συμβουλίου που θα ολοκληρώσει τρία χρόνια σε, ορισμένες, σε λίγες μέρες θα πρέπει να αναθεωρηθεί, όπως προβλέπετε, τρία χρόνια λοιπόν μετά την έγκρισή της. Αυτό λοιπόν θα μας απασχολήσει κατά τη διάρκεια του 2012. Τους τελευταίους μήνες η ΚΟΑΡΜΑ ασχολήθηκε ιδιαίτερα με, την, με τον εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη θα αναρμονίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις πολιτικές επιτήρησης των εξαγωγών όπλων και τους τελευταίους 12 μήνες προσπαθήσαμε να δραστηριοποιηθούμε ιδιαίτερα δεδομένων των όσων συμβαίνουν στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή και ασχοληθήκαμε επίσης και με τις επιπτώσεις ε, της ε, πολιτικής αυτής συγκυρίας στην πολιτική εξαγωγών όπλων των κρατών μελών. Η ε, ενώ συνεδρίαζε στο παρελθόν 9 φορές, 9 φορές για παράδειγμα το 2011 και είχε δύο άτυπες συναντήσεις που γινόντουσαν κάθε φορά από την εκάστοτε Προεδρία, αποφασίσαμε να εντείνουμε τη συχνότητα των συναντήσεών μας. Και έχουμε επίσης και έναν διάλογο με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, και με μία μη κυβερνητική οργάνωση της Βρετανίας ιδιαίτερα η οποία εξειδικεύεται στην εξαγωγή συμβατικών όπλων. Η ανταλλαγή απόψεων στα πλαίσια της ΚΟΑΡΜΑ για συγκεκριμένα ζητήματα όσον αφορά κυρίως τους πιο ευαίσθητους προορισμούς, ένα ζήτημα το οποίο συζητάμε όλο και περισσότερο στο παρελθόν. Κάθε μήνα ανταλλάγουμε, απο, ανταλλάσσουμε απόψε όσον αφορά την πολιτική εξαγωγών των κρατών μελών για τα συμβατικά όπλα και ασχολούμεθα επίσης και με τα περιοριστικά μέτρα τα οποία εγκρίνονται τόσο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης πρέπει να σας πω ότι η συζήτηση έχει δύο πτυχές. Από τη μια επικεντρωνόμαστε στο πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Τις περισσότερες φορές ή τουλάχιστον κάποιες φορές ορισμένα κράτη-μέλη δεν είχαν ακόμα εφαρμόσει τα αριθμιστικά αυτά μέτρα προκειμένου να ανταποκριθούν ταχύτατα, για παράδειγμα να αναστείλουν κάποιες άδειες που είχαν δοθεί στο παρελθόν. Και αυτό σε εθνικό επίπεδο οδήγησε στο να κινητοποιηθούν διάφορε διαδικασίε προκειμένου να προσαρμοστούν οι εθνικέ νομοθεσίε, προκειμένου το εκάστοτε κράτο μέλο να μπορεί αυτόματα άμεσα να αναστέλει μια άδεια που είχε εκχωρηθεί στο παρελθόν σε τρίτο κράτο όσον αφορά εξαγωγέ όπλων. Επίση, σε εθνικό επίπεδο, πολλά κράτη-μέλη μετά από αίτημα των Εθνικών Κοινοβουλίων τους ξεκίνησαν μια επίσημη διαδικασία αναθεώρησης των εθνικών πολιτικών στον τομέα αυτό και η αναθεώρηση αυτή βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Επίσης πιστεύω ότι η διαδικασία αυτή σε ένα βαθμό θα βαρύνει και στα πλαίσια της αναθεώρησης της κοινή θέσης, η οποία θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του 2012. Αυτά όσον αφορά την καθημερινή εργασία της ΚΟΑΡΜΑ. Θα έλεγα ότι δεν ήταν ένα συνήθις, αλλά ένας ιδιαίτερος χρόνος για την ΚΟΑΡΜΑ το 2011, γιατί η πιο σημαντική πτυχή της εργασίας μας, αυτή η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, σαφώς έλαβε χώρα αλλά έπρεπε να γίνουν και κάποιες προπαρασκευαστικές εργασίες για την αναθεώρηση της κοινή θέσης. Σύμφωνα με το άρθρο 15 της κοινή θέσης, η διαδικασία αυτή προβλέπει να ξεκινήσει σε λίγες εβδομάδες και θα μας απασχολήσει κατά το μέγιστο τμήμα του 2012 και θα πρέπει βέβαια να γνωρίζουμε ποιο είναι ο βαθμό εφαρμογή τη κοινή θέση στα κράτη-μέλη και πρέπει να δούμε αν ε, αυτή η κοινή θέση εξακολουθεί να είναι το καλύτερο δυνατό μέσο για τη ρύθμιση των εξαγωγών συμβατικών όπλων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2011 γίνανε κάποιες προπαρασκευαστικές διεργασίες, άρχισαν τα κράτη-μέλη να προετοιμάζουν τι προτάσει του για τη νέα κοινή θέση. Το όλο εγχείρημα αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ΚΟΑΡΜΑ. Κάθε κράτος μέλος εξετάζει την κοινή θέση, κάνοντας προτάσεις, αλλά περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι οι ευκαιρίες που θα έχουμε να συνομιλήσουμε όχι μόνο με τα κράτη-μέλη, αλλά και με άλλα εμπλεκόμενα μέρη όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για μία αναθεώρηση, επομένως θα γίνει ουσιαστικά μία αξιολόγηση, ένας απολογισμός του τι έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής Ξέρετε ότι έχουμε ένα νέο ουσιαστικά μέσο μπροστά μας, είναι μόνο τριών ετών και εφαρμόζεται λοιπόν αυτή η κοινή θέση τα τελευταία τρία χρόνια. Δεν έχουμε ακόμα μια παγιωμένη θέση όσον αφορά την εφαρμογή της και μια παγιωμένη αξιολόγησή της. Αποτελεί συνέχεια του κώδικα συμπεριφοράς και ουσιαστικά αποτέλεσε μια βαθμιαία διαδικασία που οδήγησε στην έγκριση αυτού του νομικού μέσου. Πρόκειται όμως ακόμα για ένα έγγραφο το οποίο είναι σχετικά πρόσφατο. Και θα πρέπει να δούμε και ποια την εφαρμογή του, ποια μαθήματα μπορούμε να αποκομίσουμε, ποια διδάγματα μπορούμε να αποκομίσουμε από την εφαρμογή του μέσου αυτού. Καταλαβαίνετε, διδάγματα αυτά θα είναι κάπως περιορισμένα στο εύρος τους. και θα πρέπει να δούμε και ποια ανάλυση θα πρέπει να κάνουμε στα πλαίσια της γενικότερης αναθεώρησης του κειμένου. Θα είναι μια διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του κειμένου, μια ανοιχτή διαδικασία η οποία θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να εντοπίσουμε και τα μέτρα εκείνα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε μια γενικότερη αναθεώρηση του κειμένου, αλλά πιστεύω ότι μάλλον θα οδηγήσει περισσότερο σε επικαιροποίηση συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν καλύτερα την κοινή αυτή θέση. Για παράδειγμα, ποιε ήταν οι παράμετροι που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να εφαρμοστεί η κοινοτική αυτή κοινή θέση. Στη φάση αυτή θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εξετάσουν την τελευταία εκδοχή του οδηγού χρήσης και να δούνε πώς θα πρέπει να τροποποιηθεί ή να επικαιροποιηθεί μετά διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει με την αναθεώρηση της κοινή θέση. Μπορώ όμως να δώσω περισσότερα στοιχεία αυτά, απαντώντας και σε ενδεχόμενες ερωτήσεις σας. Να αναφερθώ τώρα στην δεύτερη σημαντική προτεραιότητα, στην οποία θα δραστηριοποιηθεί το 2012 η ΚΟΑΡΜΑ. Πρόκειται για την διαδικασία διαπραγμάτευσης της συνθήκης για την εμπορία όπλων. Ήδη από το 2010 ξέρετε ότι μία ad hoc υποεπιτροπή της ΚΟΑΡΜ και της ΚΟΥΝΤΟΥΝ που είναι η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τον Αφοπλισμό και τον Έλεγχο των Εξοπλισμών. Μια υποεπιτροπή λοιπόν ΚΟΑΡΜ ΚΟΝΤΟΥΝ δημιουργήθηκε προκειμένου να συντονίσει την κοινή θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συνδιάσκεψη που θα γίνει. Συζητάμε μία φορά το μήνα, συνεδράζει μία φορά το μήνα η υποεπιτροπή αυτή και προσπαθούμε να διαμορφώσουμε την κοινοτική θέση σε σχέση με την μελλοντική NTT. Έχουμε κάποιες εσωτερικές κατευθύνε γραμμές και κάποια εσωτερικά έγγραφα ιδιαίτερα χρήσιμα, προκειμένου να καθοδηγήσουν τόσο την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και την παρέμβαση των επιμέρους κρατών μελών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής της διάσκεψης για την συνθήκη. Θα πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια της συνθήκης ATT η σύσταση η οποία θα δοθεί από την Προπαρασκευαστική Επιτροπή που είχε συνεδριάσει και κατά τη διάρκεια του 2010 και του 2011 και θα συνεδριάσουμε και μεταξύ, μάλλον μεταξύ 13 και 17 Φεβρουαρίου προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά το περιεχόμενο της συνθήκης. Τώρα έχουμε ένα σχέδιο κειμένου που έχει εκπονήσει ο πρόεδρος αυτής της Προσκευαστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος Μολτάν από την Αργεντινή και έχουμε συμμετάσχει και σε διμερείς επαφές και με τον Πρόεδρο και με την Προπροσκευαστική Επιτροπή και με άλλες αντιπροσωπείες για να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το κείμενο αναφοράς βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ATT και συνεχίζουμε να είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε μια εύρωστη ATT μια ισχυρή ATT με διάφορες αξιόπιστες παραμέτρους και κριτήρια που πραγματικά θα καταστήσει την εμπορία στα συμβατικά όπλα πιο διαφανή ε, και για μας ε, το 2012 είναι το τελικό αποτελέσμα που στοχεύουμε δηλαδή τον Ιούλιο του 2012 να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ε, δεν είμαστε θετικοί απέναντι στην προοπτική να ξεπεράσουμε αυτή την προθεσμία, αυτή την ημερομηνία, γιατί θεωρούμε ότι ο Πρόεδρος Μεροντάν και η Προπροσκευαστική Επιτροπή έχουν διατηρήσει την όθηση. Οι κύριοι stakeholders υποστηρίζουν αυτή τη διαδικασία. Οι ΗΠΑ το 2009 άλλαξε άποψη. Η Κίνα είναι ε, ε, ουσιαστικά πιο θετική τώρα απέναντι σε μια δεσμευτική συνθήκη, κάτι που δεν θα σκέφτονταν καν πριν ένα χρόνο και η Ρωσία φαίνεται να δείχνει κάποια δείγματα προς μετακίνηση και έτσι λοιπόν ε, είμαστε ένα μεταξύ των 50 που ψηφίσαν θετικά στον ΟΗΕ για την δεσμευτική ATT και νομίζω ότι ε, έχουμε ε, αφιερώσει και ενέργεια προς τρίτες χώρες αλλά και προς ε, τη βιομηχανία για να είμαστε σίγουροι ότι όσο και περισσότεροι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και ότι πραγματικά θα πετύχουμε στο να δημιουργήσουμε ένα μέσο που θα θέτει ίσους κανόνες στον τομέα των εξαγωγών των συμβατικών όπλων. Να σας αναφέρω και κάποιες άλλες δραστηριότητες που είναι επίσης σημαντικές για την ΚΟΑΡΜ αλλά ίσως ε, να μην είναι τόσο ε, σε σημαντικές επίπεδα. Έχουμε κάποιες δραστηριότητες για την προώθηση των κριτηρίων της κοινή θέση για τις όμορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε την, την απόφαση του Συμβουλίου που υιοθετήθηκε το 2010, 2010 κάθετος 10-12 ε, υπό την ΚΕΠΑ όπου εκεί οργανώνουμε διάφορες εκδηλώσεις κυρίως στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Νότια Ευρώπη αλλά και στο Νότιο Κάφκασο και προωθούμε την ε, κοινή θέση και φυσικά τα κριτήρια της ε, κοινή θέση. Επίσης, ε, δυνάμει αυτής της απόφασης του Συμβουλίου έχουμε σχεδιάσει κάποιες επισκέψεις ε, μελέτης, έτσι ώστε κάποιοι αξιωματούχοι από τις χώρες αυτές θα μπορέσουν να επισκεφθούν περισσότερα από ένα, μάλλον ή περισσότερα κράτη-μέλη και να δουν πώς λειτουργεί το δικό μας σύστημα εξαγωγής όπλων και εκεί μπορούν να συμμετέχουν τελειωνιακοί αξιωματούχοι, μέχρι ε, και αστυνομικοί και υπάλληλοι το Υπουργείο Εξωτερικών ή του Υπουργείου Άμυνα. Ε, έχουμε και μία επίσκεψη που θα λάβει η χώρα στην Τσεχική Δημοκρατία το 2012. Και με αυτή την τελική επίσκεψη θα ολοκληρωθεί η εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου και ήδη τώρα αξιολογούμε τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα και να σκεφτούμε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Δηλαδή ε, αυτό που αναμένουμε το είναι ότι θα έχουμε και μία νέα απόφαση ε, του Συμβουλίου για τις εξωτερικές δραστηριότητες ε, στις όμορες χώρες. Επίσης, είμαστε πολύ απασχολημένοι αυτή την περίοδο με το να διασφαλίσουμε ε, την δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης για τις εξαγωγές των συμβατικών όπλων. Ε, πρόκειται για ένα τεράστιο έργο. Ε, η έκθεση είναι 130 σελίδες ε, και δείχνει όλες τις εξαγωγέ των κρατών μελών το 2010 που εγκρίθηκαν από τα κράτη-μέλη το 2010 και πραγματικά χρειάστηκε πολύ χρόνο να εκπονήσουμε την έκθεση αυτή και ελπίζουμε μέχρι τέλη του έτους να μπορέσουμε να τη δημοσιεύσουμε. Ευχαριστώ να αναφερθώ και σε άλλε δραστηριότητε της ΚΟΑΡΜΑ εκεί όπου ήμασταν ιδιαίτερα ενεργοί, κυρίως στον πολιτικό διάλογο με τρίτες χώρες. Ε, ε, νομίζω βέβαια ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να αναφερθώ σε αυτές τις περαιτέρω δραστηριότητες, αλλά καλό είναι επομένως να σταματήσω εδώ και να ακούσω κάποιες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος έχει ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε εδώ. γιατί είμαι ένας από τους βουλευτές ε, που παρακολουθούμε το θέμα αυτό εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Και από τότε που ε, εγκρίθηκε η θέση του Συμβουλίου και έκτοτε δεν είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με την ΚΟΑΡΜ. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν καταρχήν διότι βρίσκεστε εδώ και για δεύτερον διότι έχετε ένα είδος ε, μόνιμου ρόλου στην ΚΟΑΡΜ. Οι συμφωνίες που είχαμε υπογράψει στο παρελθόν ήταν κάτι που άλλαζε, γιατί επειδή κάθε έξι μήνες άλλαζε η Προεδρία, μπορούσαμε δύσκολα να το παρακολουθήσουμε αυτά που συνέβαιναν. Μέχρι τώρα η συνεργασία μας με την ΚΟΑΡΜ πάντως ήταν πολύ επικοδομητική. Για τα θέματα τα οποία αναφέρατε, και θέλω απλώς δύο-τρία να επισημάνω από αυτά που είπατε, από το γενικότερο πλαίσιο το οποίο παρουσιάσατε έχω ένα σημείο τα προβλήματα τα οποία φαίνονται όχι για την ύπαρξη κοινή θέση, αλλά για την υλοποίηση της κοινή θέση. Ένα από τα προβλήματα έχει σχέση με το ότι συνήθως τα κράτη-μέλη προσπαθούν να κάνουν μια αξιολόγηση των μέτρων που έχουν λάβει και δεν αναλύουν την ήδη υφιστάμενη νομοθεσία, ούτω ώστε η κοινή θέση να μπορέσει να υλοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουν τα μεμονωμένα στοιχεία, το μεμονωμένο πλαίσιο κάθε κράτους μέλους, για να είναι πιο εύκολη η υλοποίηση. Ξέρουμε ότι η κοινή θέση είναι μια κοινή θέση, αλλά τα μεμονωμένα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές επιμέρους καταστάσεις, διαφορετικές βέλτιστες πρακτικές, θα έλεγε κανείς. Και θα ήθελα να ακούσουμε τι, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Συνήθως από την πείρα μου εγώ έχω δει ότι η κοινή θέση βασίζεται στον πιο χαμηλό παρονομαστή, αντί να περάσουμε στις υψηλότερες προδιαγραφές που έχουν τα κράτη-μέλη. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι θα ήταν χρήσιμο να προσανατολιστούμε προς κάτι το κοινό. Ένα δεύτερο σημείο τώρα, που έχει σχέση με την εμπειρία μας από έλεγχο. Καλό είναι να έχουμε καλή νομοθεσία. Αλλά βλέπουμε ότι μερικές φορές ε, μπορεί να υπάρχει έλλειψη ελέγχου στα σύνορα. Και η υλοποίηση της κοινή θέσης ε, θα κάνει αυτή την κατάσταση πιο πολύπλοκη. Ένα τρίτο σημείο. Η αναθεώρηση αυτής της κοινή θέσης Τι χρονοδιάγραμμα προβλέπετε για την αναθεώρηση. Ποια είναι τα προγραμματισμένα βήματα για να μπορούμε και εμείς να παρακολουθούμε τις συζητήσεις. Και ποιο είναι το πεδίο. Είπατε ότι θα είναι στενό το πεδίο, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για την αναθεώρηση, παραδείγματος χάρη η όρη συγγραφής υποχρεώσεων. Και τέλος, αν συνδυάσουμε αυτήν την αναθεώρηση με το ATT e που αναφέρατε, συμφωνώ ότι η υφιστάμενη κατάσταση στις συζητήσεις ATT ε, e φαίνονται αισιόδοξε Βέβαια, λαμβάνοντα υπόψη τι δεν έχει γίνει τα τελευταία 50 χρόνια, δεν είμαστε τόσο αισιόδοξοι. Αυτό που έχω κατά νου είναι ότι δεν, δεν πρέπει να περιμένουμε τους άλλους να πάρουν μια απόφαση. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγετική θέση στις συζητήσεις ATT και τι χρονοδιάγραμμα, τι πρόγραμμα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις συζητήσεις αυτές. Ξέρουμε πάντοτε ότι αν οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ρωσία ή η Κίνα δεν συμμετέχουν θα είναι δύσκολο. Αλλά παρόλα αυτά θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ηγετικό ρόλο σε πολλά από αυτά τα θέματα. Όλο τελικά μας λέτε, λέει ο Πρόεδρος, αλλά δεν τελειώνεται. Ε, μα δεν είναι ενδιαφέρον αυτό το θέμα, ποτέ δεν το συζητάμε. Τελευταίο, αλλά πραγματικά τελευταίο σημείο τώρα. οι, Ευρω... οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι μπορούν να κάνουν. Η έκθεση η που έχουμε τώρα ε, ενώπιόν μας μας δείχνει ότι υπάρχουν πολλά κενά όταν προσπαθούμε να έχουμε κοινή θέση. Γι' αυτό έχω την ερώτηση μου αν με βάση την εμπειρία μας από το παρελθόν ή την κοινή θέση μπορούμε να κάνουμε κάτι σε σχέση με τον κατάλογο των χωρών. Ευχαριστώ. Κυρία Λιούζιν και μετά κύριος ε, Κάμπελ. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω άμεσα ε, μετά από αυτό που είπε ο προηγούμενος ομιλητής. Κατά τη γνώμη μου, δεν τίθεται απλώς ε, θέμα ελέγχου στα σύνορα, αλλά σαφώς τίθεται θέμα εγκρίσεων και αδειών. Βλέποντας τα κριτήρια δεν θα τα παραθέσω όλα, διεθνές δίκαιο, παραβίαση, παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, εσωτερική καταστολή. Αν τα συγκρίνω όλα αυτά και βλέπω ότι τα τελευταία δέκα χρόνια στη Σαουδική Αραβία μόνο μία φορά βλέπουμε άρνηση άδειας, και το 7,2 των εξαγωγών της ε, εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνουν προς τη Σαουδική Αραβία και μόνο μία φορά αρνηθήκαμε με την άδεια ε, την έγκριση. Παρά τον κατάλογο των κριτηρίων φαίνεται ότι οι άδειε συνεχίζουν να ε, δίδονται. Τι να πούμε τώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σαουδική Αραβία τα ίδια, θα μπορούσε να πει κανείς και για τον Μπαχρέιν και άλλες χώρες. Πώς ε, βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση στο μέλλον. Θα τηρούνται τα κριτήρια για την ε, εκχώρηση αδειών. Και βλέποντας και τις περιοχές της Βορείου Αφρικής, την τελευταία δεκαετία ο ρυθμιστικός μηχανισμός υπήρχε και μας είναι γνωστό τι έχει γίνει στις χώρες αυτές. Είναι οι προτιμόμενες χώρες εξαγωγών εξοπλισμού της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό θέτω την ερώτησή μου. Και άλλη μια ερώτηση. το ότι η Γαλλία έδινε όπλα στους επαναστάτες στη Λιβύη ενώ υπήρχε εμπάργο όπλων κατά τον πόλεμο στη Λιβύη, πώς το κρίνετε. Βλέπω ότι υπάρχουν κενά όσον αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών εξοπλισμού Υπάρχουν σαφώς κενά στην οδηγία. και δεν μπορεί οι, οι ίδιες οι να συντάσσουν τις εκθέσεις. Θα είχε νόημα να υπάρχει ένας εσωτερικός έλεγχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και όχι οι εταιρείε ε, κατασκευαστών να κάνουν τις δηλώσεις. Αυτά. Ευχαριστώ. Campbell, Ευχαριστούμε κύριο Σκάμπελ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση στον κύριο Πιάτσα όσον αφορά τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Ποια δυνατότητα θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταματήσει την εξαγωγή όπλων. Θα μιλάμε ουσιαστικά για ευρωπαϊκές άδειες εξαγωγής ή για εθνικές άδειες εξαγωγής όπως γίνεται τώρα. Και η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται από ποιον, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Συμβούλιο. Και θα συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνα στα πλαίσια της συναπόφασης. Σε ποια φάση εμείς θα επεμβαίνουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητάμε, να ψηφίζουμε. Έχουν προκαθοριστεί όλα αυτά τα πράγματα, έχουν αποφασιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Διστάζω για το να σας πω να εσείς ε, συνεργάζεστε με το ΣΥΠΡΙ γιατί ξέρω ότι για πολύ καιρό ε, τηρούν ένα αρχείο για τις μεταφορές των όπλων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αν δεν σας πειράζει να ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση, γιατί νομίζω ότι αυτό όπως αφηνίζει και τις λοιπές ερωτήσεις που τέθηκαν. Δεν ξέρω αν ρωτήσετε εμένα προσωπικά, δηλαδή τι αρμοδιότητες έχουμε για να σταματήσουμε μια διεξαγωγή, γιατί να σας πω εν αυτή η ερώτηση καμία. Γιατί η απόφαση για το αν ε, θα δοθεί άδεια για μία μεταφορά, αυτό είναι αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Έτσι λοιπόν η κοινή θέση θέτει κοινά κριτήρια που κάθε κράτος μέλος ε, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όταν εξετάζει τις αιτήσει ε, για την αδειοδότηση, αλλά την τελική απόφαση την έχει το κράτος μέλος όπου έχει κατατεθεί η αίτηση. Έτσι λοιπόν αυτό δεν σημαίνει τώρα ότι τα κράτη-μέλη μπορούν ε, απλώς στη διαδικασία τους ε, απλώς να έχουν την εξέταση των παραμέτρων και εκεί βάζουμε τελεία. Υπάρχει υποχρέωση στο κείμενο στο, τις κοινής θέσης στο άρθρο 7 να, εξετάσου, να, υπάρχει, να εξεταστεί το θέμα της εναρμόνισης των πολιτικών των κρατών μελών σε αυτό το τομέα και τέτοια αποτελέσματα μπορούσαν να, να επιτευχθούν και μέσω συγκεκριμένου μηχανισμού ε, μέσα σε αυτόν υπάρχει και η ανταλλαγή πληροφοριών της ΚΟΑΡΜΑ αποτελεί ένα στοιχείο αυτού του μηχανισμού και επίσης ο μηχανισμός ε, άρνησης ανταλλαγής είναι κάτι πολύ σημαντικό για να διασφαλίσουμε περισσότερη εναρμόνιση και συνοχή στον τομέα αυτό. Όπως ε, ξέρετε, κάθε κράτος μέλος ε, που αρνείται μία μεταφορά όπλων σε ένα στο τρίτη χώρα πρέπει να το κοινοποιήσει αυτό μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέσα σε τρεις εβδομάδες μέσω ενός ασφαλού συστήματος και οποιοδήποτε κράτος μέλος που έχει μία αίτηση άδειας εξαγωγής που είναι παρόμοια ή ουσιαστικά ταυτόσιμη με αυτή που έχει τύχει άρνηση, υποχρεούται να ε, διαβουλευτεί με το κράτος μέλος που αρνήθηκε και να λάβει την απόσφαση βάσει αυτής της διαβούλευσης και να κοινοποιήσει όλους τους ενδιαφερομένους για την τελική απόφαση που έχει ληφθεί σχετικά με το αν θα επιτραπεί όχι μεταφορά. Έτσι λοιπόν ε, αυτό είναι ένα στοιχείο που νομίζω ότι εξακολουθεί να έχει αποτελέσματα. Είναι ε, πολύ πρόημο να αξιολογήσουμε τον τελικό του αντίκτυπο. Όμως, ε, κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ελέγχου των πολιτικών των κρατών μελών. και να σας πω ότι δεν παραμένουμε στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή, γιατί αν υπάρχει ένα κρατός μέλος ε, το οποίο ε, είναι πάρα πολύ διστακτικό και αρνείται ε, πάρα πολλές μεταφορές, δημιουργεί υποχρέωση και στους υπολείπους, στα υπόλοιπα κρατημέλη, να ζητήσουν τη συμβολή του. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπα, είναι μάλλον θέμα αύξησης του πύχη εδώ. Τώρα, για να έρθω στην άλλη ερώτηση, αντίστροφα κινούμε. Σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Θα αναφερθώ στην ε, ερώτηση της κυρίας Λίζενγκ. Το πρόβλημα ότι είναι όχι μόνο με τους ελέγχους αλλά και με τις ίδιες τις εγκρίσεις, με τις ίδιες τις εγκρίσεις. Εσείς ε, είπατε ότι ε, πάρα πολλές φορές εστάλησαν όπλα σε χώρες που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ήθελα να πω ε, τρία πράγματα εδώ. Όπως ε, ανέφερα, υπάρχει υποχρεώση αξιολόγησης καταρχήν ε, που γίνεται αναπερίπτωση από κάθε κράτος μέλος για κάθε αίτηση εξαγωγής. Και τι σημαίνει αναπερίπτωση. Ότι κάθε φορά που εξελογείται μία αίτηση εξαγωγής πρέπει να δείτε τα είδη των όπλων, τι είδος όπλα εξαγεται το ποσοστό ε, που εξαγεται τον τελικό χρήστη που έχει δηλωθεί, την τελική χρήση που έχει δηλωθεί και την αξιοπιστία των πληροφοριών που σας έδωσαν. Δηλαδή, εκτός ε, και αν υπάρχει εμπάργκο δεν μπορείτε να έχετε μια χώρα στη μαύρη λίστα γιατί υπάρχουν όπλα που θα μπορούσατε υπεύθυνα να στείλετε σε μια τρίτη χώρα γνωρίζοντας ε, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα όπλα αυτά. Τώρα τα αναφέρω γενικά όλα αυτά, αν θέλετε λεπτομέρειες θα σας τις πω. Αν ε, παραδείγματος χάρη πουλήσει ε, ένα αεροσκάφος ή ένα πολεμικό πλοίο, δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό ε, για, κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φυσικά εξαρτάται και σε ποιον το πουλάζει. γιατί μπορεί να διαφέρει ο τελικός χρήστης. Έχουμε το Υπουργείο Ιστορικών, το Υπουργείο Άμυνας, έχουμε και κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις, non-state actors και κάθε φορά πρέπει να γίνεται σε αυτή τη βάση αξιολόγηση, λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την κάθε περίπτωση, δηλαδή λαμβάνουμε υπόψη τι αναφέρεται στην ίδια την αίτηση της εξαγωγής. Και τα στοιχεία που μπορεί να βρείτε στην ετήσια έκθεση βλέπετε όλα τα είδη των όπλων ανακατηγορία και βλέπετε και τις ποσότητες και τις αξίες και την αξία των όπλων που εξάγονται. Αυτό δεν αρκεί πάντοτε για να κρίνετε τι ακριβώς ε, αποστέλλετε, γιατί αν ε, δεν ξέρετε για τι πράγμα μιλάτε, είναι πολύ δύσκολο να κρίνετε. Αν κάτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά ενών των κριτηρίων που συμπεριλαμβάνονται στην κοινή θέση. Κατά παραβίαση δηλαδή των κριτηρίων αυτών. Νομίζω ότι ε, μπορεί να υπάρχει και αποτυχία αξιολόγηση από το κράτος μέλος, αλλά όπως ε, σας είπα έχουμε τις παραμέτρους και την τελική απόφαση, τι λαμβάνει το κράτος μέλος και φυσικά την ευθύνη την έχει το κράτος μέλος. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι ο μηχανισμός διαφάνειας που ε, αναπτύσσεται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας από τους πιο προηγμένους που μπορείτε να βρείτε στον κόσμο και αυξάνει την ε, ευθύνη των κρατών μελών. Γιατί όταν τα κράτη-μέλη αποφασίσουν να επιτρέψουν μια εξαγωγή, αυτό σημαίνει ότι μπορούν και να την υπερασπίσουν ε, τους λόγους για τους οποίους την ε, επέτρεψαν, γιατί ξέρουν ότι μπορεί να ελεγχθούν τα κράτη-μέλη και μάλιστα μπορεί να ελεγχθούν πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλα τρίτα κράτη που δεν δημοσιεύουν τέτοιες λεπτομερείς αιτήσεις εκθέσεις όπως εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση τώρα με τη δυνατότητα να έχουμε ελέγχους στο εσωτερικό των ίδιων των βιομηχανιών ή των επιχειρήσεων. Και όχι μόνο ex post ελέγχους, αν κατάλαβα την ερώτησή σας. Δημιουργείται ένα τέτοιο σύστημα, όχι ε, όμως απαραίτητο για Αυτέ τι εξαγωγέ δηλαδή. Θα έχουμε ένα τέτοιο σύστημα που θα ισχύει για τα 27 κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις ε, μεταφορές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκή Ένωση. και αυτό αποτελεί τμήμα τη οδηγία ACT που υιοθετήθηκε το 2009 και αφορά το εσωτερικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εθνικό επίπεδο βέβαια τα κράτη-μέλη έχουν ε, καθιερωμένες πρακτικές για να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν μέτρα ελέγχου και πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις τους. Αυτό ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία. Τώρα, για να έλθω στις ερωτήσεις ε, που τέθηκαν. Από τον κύριο Ρωμέβα για τα προβλήματα με την εφαρμογή και την έλλειψη νομικής ανάλυσης των όσων γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Όπω είπα, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν σε όσα συμπεριλαμβάνονται στην κοινή θέση, σε τίποτα λιγότερο, σε τίποτα περισσότερο. Επίση, συμφώνησαν να αναπτύξουν έναν οδηγό χρηστών, που είναι ένα πολιτικά δεσμευτικό έγγραφο, όπου έχουμε κατευθύνε γραμμέ και βέλτιστε πρακτικέ και επικαιροποιείται και συχνά το έγγραφο. Αυτό είναι το αποτελέσμα τη ε, αναθεώρηση τη κοινή θέση, που αναμένω να προκύψει, είναι ότι θα έχουμε μια ουσιαστική αναθεώρηση και επικαιροποίηση αυτού του οδηγού. Εκεί θα έχουμε κατευθυντήρες γραμμές για το πώς ερμηνεύονται οι παράμετροι, πώς ε, αξιολογούμε μία αίτηση, ε, πώς ε, προσδιορίζουμε να έχουμε ταυτόσιμες συναλλαγές. Έτσι λοιπόν υπάρχει δυνατότητα να δούμε τα διδάγματα από το παρελθόν και έτσι στην αναθεώρηση του οδηγού θα έχουμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρατε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία της αναθεώρησης, δεν ήθελα να πω ότι θα είναι στενό το πεδίο ε, της αναθεώρησης. Δεν είναι αυτό το σημείο αφετηρίας. Ε, νομίζω ότι μάλλον αυτό θα είναι το σημείο αφετηρίας, γιατί θα ήταν κοντόφθαλμο να περιορίσουμε τα αποτελέσματα τα ενδυνάμει αποτελέσματα τη κοινή θέση πριν ε, να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του, του έχουμε πετύχει. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούγεται λογικό τρία χρόνια μόνο μετά την υιοθέτηση της νομικής πράξης θα ήταν ίσως πρόημο να αρχίσουμε από το μηδέν, να καταργήσουμε τα πάντα και να ξεκινήσουμε από το μηδέν και να πούμε ότι τα πάντα θα πρέπει να αναδιατυπωθούν. Και αυτό επειδή είναι περιορισμένη η εμπειρία που έχουμε συσσωρεύσει μέχρι τώρα. Αν θεωρείτε ότι ο κώδικα διοντολογία, αν σκεφτείτε ότι ο κώδικα διοντολογία ευθύθηκε το 1998 και μόλις, μετά το 2008 ψηφίστηκε η κοινή θέση, αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου και να σας πω ότι η αναθεώρηση δεν ε, είναι μια διαδικασία ε, η οποία θα τελειώσει. Είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Και ε, το 2012 θα κάνουμε και μια αποτίμηση. Τους πρώτους μηνές του 2012 φαντάζομαι ότι θα ασχολούμαστε με το εγχείρημα της ε, αξιολόγησης που ξεκινήσαμε ήδη σε σχέση με τις συγκεκριμένε ερωτήσεις που έχουν τεθεί στα κράτη-μέλη για να αξιολογήσουν τι έχουν πετύχει μέχρι τώρα και μάλλον τους επόμενους μήνες θα προβούμε σε μια ουσιαστική συζήτηση ε, του τι θα προκύψει από αυτή την αξιολόγηση και θα προσδιορίσουμε συγκεκριμένα σημεία όπου μπορεί να υπάρξει βελτίωση ή αλλαγή. Όμω ε, μπορεί τα κράτη-μέλη να μα πούν ότι είναι αρκετά ικανοποιητικά τα πράγματα όσο έχουν. Όπω σα είπα, αυτή είναι μια διαδικασία όπου τον ηγετικό ρόλο έχουν τα κράτη-μέλη, αυτά συμφώνησαν επί της κοινή θέση. αυτά θα αποφασίσουν αν αυτό το μέσο αρκεί για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ε, κατάλογο αυτών ε, των χωρών. Δεν έχουμε τέτοιο κατάλογο όπου να αναφέρουμε country of concern, δηλαδή τις χώρες που μας ανησυχούν. Ε, ίσως ε, τα κράτη-μέλη να μας το προτείνουν αυτό στη μέρα της αναθεώρησης. Ε, τώρα, τι έχουμε. Έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων για τις εξαγωγές που επιτρέπονται και που αξιολογούνται έναντι συγκεκριμένων χωρών. Και σε κάθε συνάντηση ΚΟΑΡΜΑ, από πριν μάλλον θα έλεγα, ε, αποφασίζουμε τι θα συζητήσουμε στην επόμενη συνάντηση. Αυτό δεν δημιουργεί υποχρέωση ψηλότερου ελέγχου, αλλά αν δεχτείτε το γεγονός ότι ε, ένα από τα αποτελέσματα της κοινή θέση είναι ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να διαβουλεύονται με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και να ακούν το ένα τον άλλο. Ε, αυτό το στοιχείο, δηλαδή το αν ο προορισμός των όπλων είναι ανησυχητικό, είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε. Θα πρέπει βέβαια τα κριτήρια να τα εφαρμόζουμε με αυστηρό τρόπο και φυσικά αν υπάρχουν και αποκλίνουσες απόψεις, γι' αυτό ενημερώνονται όλα τα κράτη-μέλη. Συμφωνώ ότι αυτό είναι κάτι που ουσιαστικά είναι à la carte Δηλαδή αντιδρούμε έναντι συγκεκριμένων χωρών, αλλά θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε στα πλαίσια της αναθεώρησης. Ίσως να προταθεί αυτό, δηλαδή να υπάρξει μια πιο διαρθρωμένη κωδικοποίηση του συστήματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας έχουν δώσει και 10 επιπλέον λεπτά οι διερμηνείς. Τους ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εξηγήσεις αυτές. Ευχαριστούμε και τους ε, συναδέλφους για το ενδιαφέρον που επέδειξαν. Ελπίζω ότι τώρα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα από όσα γνωρίζαμε πριν από αυτή τη συνάντηση και καλή σας τύχη.